ο Ζαν Πιέρ Γκαρσέν από τον ΩΣΑ ε, και η κυρία Εύκενς καταρχήν, η οποία άρχισε τη σταδιοδρομία της στις ε, κάτω χώρες, ε, χώρες ήταν πρέσβερας στις κάτω χώρες, ήταν υπουργό συνεργασίας και ανάπτυξης των κάτω χωρών πριν γίνει αυτό που είναι αυτή τη στιγμή ε, συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Δεν θα μακρηγορήσω περισσότερο, αλλά θα δώσω το λόγο στην κυρία Εύκενς. Um, Ευχαριστώ, θα μιλήσω αγγλικά. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για την συνοχή στην αναπτυξιακή πολιτική. Μου είπατε ποιο είναι το, το βιογραφικό μου, αλλά ήμουνα και βουλευτήνα ε, Ολλανδέζα στις αρχές δεκαετία του 80, εκείνη την εποχή που στην Ολλανδία προσπαθούσαμε να προωθήσουμε αυτή την πολιτική στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο ε, στη δεκαετία του 80. Πριν εμφανιστεί αυτή η έκφραση στην ε, συνθήκη του Μάστριχτ, ε, για πρώτη φορά αναφέρεται στη συνθήκη του Μάστριχτ αυτός ο όρος και λέγεται μάλιστα ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη να ληφθούν υπόψη οι αναπτυξιακοί στόχοι σε όλες τι πολιτικές μας, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τότε στο ε, Ολλανδικό Κοινοβούλιο ήμουνα εκπρόσωπο του κόμματός μου για θέματα ανάπτυξης και από τότε είχα συνειδητοποιήσει πόσο μάταιες ήταν αυτές οι προσπάθειες βοήθειας σε σχέση με την επίπτωση άλλων πολιτικών. Γι' αυτό λοιπόν ως βουλευτής εξόψα πολύ χρόνο και ενέργεια για να προωθήσω αυτή την συνοχή ε, υποβάλλοντας και δύο έγγραφα για την ε, χρηματοδότηση της ε, πολιτικής αυτής και την ανάπτυξη του εμπορίου που χρόνια μετά εξακολουθούν να είναι επίκαιρα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι η έλλειψη συνοχής στην στις κυβερνήσεις μας ήταν και είναι κάτι που αντικατοπτρίζεται και τη συστάση των κοινοβουλίων μας. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν ε, τα κυβερνητικά χαρτοφυλάκια. Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση έτσι γόνιμη. Και οι επιτροπές ανάπτυξης είναι κάτω-κάτω στην αλυσίδα ε, σημασία των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Δεν έχουν καθόλου ε, επιρροή και 20 χρόνια μετά τα ίδια ισχύουν. Ε, θυμάμαι ε, το ψήφισμα που πέρασε το Κοινοβούλιο για την ε, κοινή αγροτική πολιτική και για τις επιδοτήσεις. Εκείνη τη στιγμή γινόταν μια διάσκεψη παράλληλα για την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις. Εμείς ε, εκεί θα έπρεπε να είμαστε και όχι σε αυτήν εδώ τη διάσκεψη θα μιλάμε μεταξύ μας. Μια δεύτερη παρατήρηση είναι ότι το 1992 κωδικοποίησαμε αυτή την πολιτική. Ξαναμιλήσαμε το 2005 στην Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη, αλλά οι μηχανισμοί εφαρμογής δεν υπάρχουν. Ούτε και σήμερα. Και οι πολιτικές δεσμεύσεις είναι επίσης πολύ γενικές και αόριστες. Πολλά κράτη-μέλη κρύβονται πίσω από την κοινότητα και το κοινοτικό επίπεδο λένε ότι δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν κοινοτικέ δεσμεύσει. Αλλά αν δεν ε, ανασκουμποθούν και οι εθνικέ μα κυβερνήσει ε, για αυτή την συνοχή στην αναπτυξιακή πολιτική, δεν θα τα καταφέρουμε. Ορισμένα κράτη-μέλη δεν αναγνωρίζουν καν το γεγονό ότι συμφωνήσαμε ότι πρέπει να είμαστε συνεπεί και συνεκτικοί. Δεν βλέπω κανέναν Ιταλό βουλευτή. Αν δείτε όμω την ε, έκθεση τη Επιτροπή ΝΤΑΚ για την Ιταλία, δεν, υπάρχει, δεν αναφέρεται καθόλου αυτό το θέμα εκεί. Όταν έγινε λοιπόν υπουργό Αναπτυξιακή ε, Συνεργασία, ε, είναι ότι πολύ λίγα ε, κράτη-μέλη έχουν υπουργό ανάπτυξη. Και ακόμη και αν έχει, οι φωνέ των φτωχών δεν πρέπει να ακουστούν στο επίπεδο που λαμβάνονται οι αποφάσει. Και χωρί έναν πραγματικό επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίο θα είναι υπεύθυνο για όλου του πόρου τη επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, τότε η αναπτυξιακή τα αναπτυξιακά θέματα θα χάνουν ε, εις βάρος άλλων εθνικών θεμάτων που έρχονται πρώτα. Τώρα θα ήθελα να πω δύο λόγια για θέματα μετανάστευσης. Εγώ ήμουν σε αυτή την ε, κυβέρνηση η οποία το 2002 έπεσε από την εξουσία γιατί δεν έκρινε σωστά την επίπτωση της αυξανόμενης ε, μετανάστευσης από χώρες με άγνωστες κουλτούρες στη δική μας εθνική ταυτότητα, στις αξίες μας, στην κοινωνική συνοχή μας. Ε, και επίση ε, δεν κρίναμε σωστά την ικανότητα απορρόφηση ε, των μεταναστών στην κοινωνία μα. Επομένω, καταλαβαίνω τι δυσκολίε που έχουν οι πολιτικοί να μιλήσουν ανοιχτά, στεναρά. Αλλά πραγματικά είναι και καινή ώρα και, και χαίρομαι που και οι εκπρόσωποι του ΩΣΑ είπαν το ίδιο πράγμα. Είναι ώρα λοιπόν να αναλυφθούν οι ευθύνε, να γίνουν αυτέ οι συζητήσει, να υπάρξει λιγότερη ξενοφοβία. Δεν θα πρέπει να κατηγορούμε ανθρώπου λόγω τη προέλευσή του. Η μετανάστευση υπάρχει και θα παραμείνει. Και ξέρω ότι αυτή τη στιγμή μας απασχολεί οικονομική ύφεση. Βλέπουμε ότι οι Πολωνοί εργάτες φεύγουν από το Λονδίνο και το Δουβλίνο και βλέπουμε ότι οι Μεξικανοί ε, φεύγουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, βλέπουμε ότι τα εμβάσματα μειώνονται και τα 200 εκατομμύρια άνθρωποι που έφυγαν από τα σπίτια τους για να αναζητήσουν καλύτερη ζωή πραγματικά δυσκολεύονται. Ζουν ε, πολύ άσχημα σήμερα καθώς ε, υπάρχει ύφεση, καθώς ε, αυξάνεται η ανεργία και τους χτυπάει πρώτους βέβαια τους μετανάστες. Και ακόμα πολύ συχνά από πολλούς πολιτικούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να αρπάξουν τις ψήφους ε, των υπηκών τους ότι να σκληραίνουν τη γλώσσα. Κοιτάμε την, την οικονομική κρίση για τους προσπαθούμε να προωθήσουμε πακέτα για τους υπηκόους μας και ο Βρετανός ε, Πρωθυπουργό μιλάει για τις θέσεις απασχόλησης ε, για τους βρετανού υπηκόου. και με ανησυχούν πάρα πολύ όλα αυτά. Αλλά πιστεύω ότι όταν περάσει η ύφεση θα αυξηθεί η μετανάστευση. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ε, φυγόκεντρες τάσεις και κεντρομόλες τάσεις. από τη μία οι άνθρωποι πρέπει να αναζητούν ας πούμε, προσπάθειες εδώ να χτίσουν τη ζωή τους και από την άλλη και η αγορά εργασίας μας τους χρειάζεται. Όλα αυτά πρέπει να τα αναγνωρίσουμε και το έκανε και η Επίτροπο σήμερα το πρωί. Τμήμα τη οικονομία μα και των δημοσίων υπηρεσιών μα εξαρτώνται από τα ξένα εργατικά χέρια. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η δική μα εφημερία, ιδίω σε χώρε με τεράστια δημογραφικά προβλήματα εξαρτώνται πάρα πολύ από τους ε, μετανάστες. Τους χρειαζόμαστε αν θέλουμε να κρατήσουμε το επίπεδο της οικονομικής παραγωγικότητάς μας και αν θέλουμε να έχουμε τις συντάξεις μας, την κοινωνική ασφάλιση, εάν θέλουμε να μας φροντίσει κάποιος όταν γεράσουμε. Η μετανάστευση είναι μια συνέπεια, δεν είναι η αιτία ε, της έλλειψης ανάπτυξης. Ιδίως ε, και είναι και θέμα έλλειψης ευκαιριών στις χώρες προέλευσης και θα πρέπει να διατηρήσουμε τις ελάχιστες αναπτυξιακές πηγές που έχουμε για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, να, να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του, να μην διασπαθήσουμε αυτά, αυτούς τους πόρους που έχουμε, ε, προσπαθώντας να ασχοληθούμε με τα συμπτώματα. Χρειαζόμαστε συνέπεια για να προωθήσουμε τις ε, πολιτικές μετανάστευσης για την ανάπτυξη και όχι το αντίθετο. Τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ε, τιμούν τι ε, δεσμεύσει του ό,τι αφορά την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, σε ό,τι αφορά την ποιότητα και τον όγκο. Εμείς η Ευρώπη έχουμε δεσμευτεί ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη μείωση τη φτώχεια ε, για τους φτωχού ανθρώπου στι φτωχότερε χώρε, ειδικά στην Αφρική. Και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Αν τη χρησιμοποιήσουμε για να εμποδίσουμε τη μετανάστευση, και αυτό συμβαίνει σε πολλά κράτη-μέλη, αυτό δεν είναι συμβατό με που έχουμε θέσει στον εαυτό μα. Επίση, η συνοχή στην αναπτυξιακή πολιτική δεν αφορά μόνο τη μετανάστευση. Θα ήθελα να σα πω ότι οι πολιτικέ μα για το εμπόριο δεν είναι συνεπεί. Πώς μπορούμε να επιμένουμε, πώς μπορούμε να περιμένουμε ότι άνθρωποι από ξένες χώρες, από τρίτες χώρες που δεν μπορούν να χτίσουν τη ζωή του εκεί, δεν θα έρθουν εδώ προφανώ να ζητήσουν καλύτερη ζωή. Επομένω, συνοχή σημαίνει και ε, εμπορικέ πολιτικέ. Και για θέματα μετανάστευση. Στο, στο ΜΠΟΕ σήμερα το πρωί... Σήμερα το πρωί μιλήσαμε για το πολυμερέ επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει εδώ και πάνω από μια δεκαετία να έχουμε μια απελευθέρωση στι υπηρεσίε. Αν δεν εξετάσουμε τι διαπραγματεύσει ε, σε επίπεδο Γκάτσεπ στον ΠΟΕ, αν εξετάσουμε μάλλον αυτές τις διαπραγματεύσεις θα δούμε ότι στις πλούσιες χώρες δεν επιτρέπουμε την προσωρινή μετακίνηση των φυσικών προσώπων. Μόου 4 στην ΓΚΑΤΣ. Δηλαδή, υπάρχει... Μιλάμε για τις δεσμεύσεις για να ανοίξουμε ε, τις υπηρεσίες σε ξένους παρόχους. Μιλάμε για την προσωρινή μετανάστευση, ε, για να σταματήσει η διαρροή εγκεφάλων. Ε, με τρόπο ούτω ώστε οι χώρε προέλευση να υποφεληθούν από τι δεξιότητε των ανθρώπων που επιστρέφουν στι χώρε αυτέ λόγω τη κυκλική μετανάστευση. Η προσωρινή μετανάστευση επίση θα αυξήσει τα εμβάσματα. Γιατί όταν κάποιο μένει πολύ α, καιρό μακριά από την πατρίδα του, μειώνεται τα εμβάσματα. Οι αναπτυγμένε χώρε όμω και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τη φιλελευθερωποίηση την ε, συνδέουμε με τον Mode 3. Δηλαδή ουσιαστικά με το πώ θα λειτουργούν οι δικέ μα τράπεζε εκεί, στι αναπτυσσόμενε χώρε. Αυτό φυσικά δεν είναι προ το συμφέρον των φτωχών χωρών, γιατί αυτό το είδο μετανάστευση ε, αφορά μόνο πολύ καταρτισμένου ανθρώπου, ε, προσωπικό μεγάλων εταιριών που πηγαίνουν σε αυτέ τι χώρε για να δουλέψουν. Κάτι άλλο που θα έπρεπε να κάνουμε είναι οι συντάξει να μπορούν να μεταφέρονται από χώρα σε χώρα, οι μετανάστε να μπορούν να τι μεταφέρουν δηλαδή να τους επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Επίσης, οι πολιτικές μας υγείας δεν είναι συνεπείς με τις πολιτικές μετανάστευσης. Νομίζω θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο εμείς οι ίδιοι για να καταρτήσουμε εμείς γιατρούς και νοσοκόμες για να φροντίσουμε τους ηλικιωμένους. Γιατί είναι απαράδεκτο ότι οι γιατροί από το Μαλάουι ε, δουλεύουν ε, πιο πολύ στο Μάντσεστερ από το στο Μαλάουι τα συστήματα υγείας εξαρτώνται όλο και περισσότερο από νοσοκόμες, γιατρούς, από την Αφρική. Και χρησιμοποιούμε την ελάχιστη ε, αναπτυξιακή βοήθεια που έχουμε και να στείλουμε μεγάλους γιατρούς πίσω στην Αφρική. Στο παρελθόν, αν δίναμε αυτά τα λεφτά στα Υπουργεία Υγείας στην Αφρική, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνητρα για να κρατήσουν δεκάδες χιλιάδων ε, γιατρούς ε, εκεί και να μην φύγουν. Κάτι που είναι σημαντικό και το είπε ο εκπρόσωπος του ΟΣΑ σήμερα το πρωί είναι ότι η μετανάστευση ουσιαστικά βοηθάει τις αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Κεντρική Αμερική, στο Πακιστάν, τα εμβάσματα ε, πληρώνουν ε, για να, σταλούν τα παιδιά στο, να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Επιτρέπει στις, μητρέ, στις μητέρες όταν γεννάνε να βοηθηθούν από ένα γιατρό κτλ. Επομένως έχουμε θετικές επιπτώσεις. Τα εμβάσματα δηλαδή ε, συντελούν στην επίτευξη των στόχων. Αλλά και το πιο σημαντικό που θέλω να πω είναι το εξή. Είναι το εξής. Στι φτωχέ χώρε δεν επωφελούνται κυρίω οι φτωχοί άνθρωποι. Το 2007 οι 10 πιο σημαντικέ χώρε, 5 μάλλον, Ινδία, Κίνα, Μεξικό, Φιλιππίνες, Γαλλία, είναι αυτέ που υποφελήθηκαν περισσότερο από τα εμβάσματα. Και είναι αλήθεια ότι τα εμβάσματα είναι τριπλάσια από τη βοήθεια. Αλλά αυτό δεν αφορά την ε, υποσαχάρη Αφρική. Στην υποσαχάρη Αφρική η μετανάστευση είναι εσωτερική και παίρνει μόνο το 2% των συνολικών παγκόσμιων εμβασμάτων. Τα εμβάσματα είναι ιδιωτικά κονδύλια. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις δημόσιες υπηρεσίες, για επενδύσεις τις οποίες τις χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Οι μετανάστες ουσιαστικά ε, είναι οι άνθρωποι που μπορούν να φύγουν από τη χώρα τους. Δεν είναι οι πιο φτωχοί, γιατί οι πιο φτωχοί δεν μπορούν να φύγουν. Επίσης, με ανησυχεί η πρωτοβουλία για την μπλε κάρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα δυσκολέψει τα πράγματα. Θα βοηθήσει μόνο αυτούς που έχουν προσόντα ήδη. Και πραγματικά αυτό δεν βοηθάει την ανάπτυξη. Τώρα, θα ήθελα να καταλήξω ότι σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο με μεγάλη κίνηση των κεφαλαίων αγαθών και υπηρεσιών ο κόσμος έχει κολλήσει κάπου. Εκτός κι αν είσαι καταπληκτικός, α πούμε γιατρό, ε, ειδικό σε θέματα ε, ε, νέων, τεχνολογιών, νέων τεχνολογιών κτλ. Τους μετανάστες όμως κανένας δεν τους κοιτάει. Θα πρέπει να σπάσουμε τα εμπόδια, θα πρέπει να δημιουργήσουμε γέφυρες. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα πολυμερές πλαίσιο. Θα πρέπει να διαχειριστούμε σωστά την μετανάστευση. Εγώ ήμουν μέλο τη επιτροπή για τι κοινωνικέ επιπτώσει τη παγκοσμιοποίηση. Και μία από τις ιδέες που είχαμε πριν από πέντε χρόνια ήταν ακριβώς αυτή. Αλλά δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα έκτοτε. Θα έπρεπε να επιστρέψουμε γύρω από μια απο τι ιδέε που ειχαμε πριν απο πεντε χρονια ηταν ακριβώ αυτη αλλα δεν τράπεζα και να δούμε πώ θα υλοποιήσουμε αυτό το πολυμερέ επίπεδο. Αυτό θα μα βοηθούσε και εμά τι βιομηχανικές χώρε που ε, έχουμε προβλήματα εκδημοκρατισμού αλλά και τι χώρε προέλευση των μεταναστών Πέντε χρόνια μετά από την διατύπωση αυτής της ιδέας δεν υπάρχει ακόμα αυτό το πολυμερές επίπεδο. Πρέπει να το δημιουργήσουμε. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε πραγματικά. Ε, γιατί δεν θέλουμε άλλες διασκέψεις. Δεν θέλουμε άλλες διασκέψεις, θέλουμε δράση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Σκέντς για την σαφέστατη και στρατευμένη παρέμβασή σας. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Καρτσόν, ο οποίος ε, ε, ε, δουλεύει για τον ΟΣΑ και που έκανε την τελευταία ε, έκθεση για τη μετανάστευση. Έχει το λόγο. Κύριε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου τιμή που μπορώ να παρουσιάσω αυτή την, ε, την ομιλία μου ε, εδώ. Ε, κατά τη διάρκεια του φαγητού είχα την ευκαιρία, όπως του μπουφέ, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με πολλούς που πραγματικά εξεπλάγησαν με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο ΩΣΑ στον τομέα της ανάπτυξης και της μετανάστευσης. Συχνά όσα είναι γνωστό σαν μια, ένας οικονομικός οργανισμός, μάλλον στην απελευθέρωση κλπ. Αλλά είναι ένας οργανισμός ο οποίος εργάζεται από την εποχή της ίδρυσής του με αναπτυξιακά θέματα και έχουμε μια λέσχη η οποία προσανατολίζει τις αφρικανικές χώρες και στο εσωτερικό του οργανισμού έχουμε μια ένωση που ασχολείται με θέματα μετανάστευση και η οποία καταρτίζει ετήσιες εκθέσει σε θέματα μετανάστευση. Αλλά υπάρχουν επίση και πολλέ άλλε εργασίε, στο επίπεδο τη μετανάστευση και τη ανάπτυξη. Σήμερα το θέμα το οποίο τίθεται από την άποψη εκείνων που ενδιαφέρονται ιδιαίτερω για το θέμα τη ε, μετανάστευση και προσπαθούν να κάνουν μια γέφυρα με την ανάπτυξη είναι κατά πόσο η μετανάστευση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Μα είπαν ναι, με, μέσω ορισμένων στοιχείων, μεταφορά ε, πόρων, εμβάσματα κλπ. Μπορεί να υποβοθεί στην ανάπτυξη. Αλλά αν ήταν μόνο η μετανάστευση, εδώ και πολύ καιρό πολλές χώρες που είναι χώρες μετανάστευσης θα έπρεπε να είχαν αναπτυχθεί. Άρα δεν αρκεί. Και παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα παραδείγματα. Σήμερα το πρωί ακούσαμε το παράδειγμα της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και επίσης της Ιταλίας Α πούμε, ο Λιμπατσί, ο οποίος είναι μεγάλος γνώστης αυτών των θεμάτων. Και θα ήθελα να πω ότι πράγματι στην Ευρώπη έχουμε χώρες όπως η Ιλλανδία που είναι μεγάλε χώρε μετανάστευση και που εδώ και κάποιε κάποιες χώρες αποστέλουν μετανάστες. Ε, δέχονται συγγνώμη μετανάστες. Ε, επίσης έχουμε τα διαφορετικά ταμεία τη Ευρωπαϊκής Ένωση, που είναι ιδιαίτερο σημαντικά και τα οποία επέτρεψαν την ανάπτυξη της Πορτογαλίας, τη Ελλάδα κλπ. Πιστεύω λοιπόν ότι η μετανάστευση μπορεί να βοηθήσει, αλλά πρέπει να υποβοηθήσουμε τη μετανάστευση, ώστε να μπορεί να έχει μια επίπτωση στην ανάπτυξη. Τώρα, το θέμα τη μετανάστευση, όπω το είδαμε σήμερα το πρωί με τόσε παρεμβάσει σε σχέση με την κρίση, είναι ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται στην καρδιά των πολιτικών συζητήσεων, στην καρδιά της γεωπολιτικής επίσης και κάποιων ε, θεμελιωδών ανθρώπινων διαστάσεων. Δηλαδή μπορούμε να προσπαθήσουμε να εμποδίσουμε τους ανθρώπους να εισέρχονται στις χώρες, τουλάχιστον να επιβραδύνουμε αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ δύσκολο να τους ξαναστείλουμε πίσω, να τους ζητήσουμε, να τους αναγκάσουμε να επανεπατριστούν. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα, αλλά είναι ιδιαίτερως περιορισμένα. Είναι πολύ δύσκολο να υποχρεώσουμε ε, τους ανθρώπους να επαναπατριστούν. Συνεπώς λοιπόν το θέμα αυτό δεν, είναι, δεν αφορά εμπορεύματα, αλλά ανθρώπινα όντα με τις οικογένειές του και υπάρχουν πολλαπλά κοινωνικά και πολιτικά διακυβεύματα. Επίσης υπάρχει ένα, είναι ένα θέμα το οποίο υποκρύπτει μεγάλη υποκρισία. Ε, μιλάμε πολύ για την ε, φυγή των εγκεφάλων, για το brain drain, και... αλλά ε, τουλάχιστον στη δική μου διεύθυνση εδώ και πολλά χρόνια παρακολουθούμε τις μεταναστευτικές πολιτικές και μπορώ να σας πω ότι τη τελευταία δεκαετία τα πιο σημαντικά μέτρα τα οποία λήφθησαν όσον αφορά τη μετανάστευση είναι μέτρα για να προσελκυστούν ειδικευμένοι εργαζόμενοι, εργαζόμενοι με ψηλά προσόντα, για να δοθούν κίνητρα ε, σε πολλού φοιτητέ, ούτω ώστε να εργαστούν σε κάποιε χώρε μετά τι σπουδέ του. Και από την άλλη, οι χώρε από τι οποίε προέρχονται αυτή η μετανάστευση δεν έχουν πάντοτε τι πολιτικέ για να μπορέσουν να κρατήσουν αυτά τα ειδικευμένα, τα εξειδικευμένα άτομα, τους δώσουν ε, τις δυνατότητες να χρησιμοποιήσουν τα προσόντα τους. Συνεπώς όλη αυτή η συζήτηση για το brain drain κλπ. είναι μια συζήτηση που θα έπρεπε καταρχήν να διευκρινίσει να διαλευκανθεί. Δηλαδή από τη μία να δημοσιευθούν στατιστικά στοιχεία για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε σε αυτό το τομέα και αυτό είναι ο ρόλος του ΟΣΑ και στον τομέα της υγείας. Εδώ υπάρχουν στατιστικές που αναφέρθησαν σήμερα το πρωί και μπορούμε να τις αναφέρουμε γιατί έχουν γίνει εργασίε σε σχέση με την απασχόληση κλπ. Για να δούμε ποιοι είναι οι μετανάστες, σε ποιους τομείς, σε ποιους κλάδους δουλεύουν, πότε ήρθαν σε λόγο χώρα, πού είναι, υπάρχει μεγαλύτερη πυκνότητα, μεγαλύτερη συγκέντρωση μεταναστών ε, και ποιο είναι το επίπεδο εξειδικευσής του κλπ. Αυτό μπορεί να μας κάνει να ε, κάνουμε την προβληματική αυτή κάπως πιο ακριβή. Τώρα, το άλλο θέμα είναι το θέμα της δημογραφίας. Βγαίνονται ε, σχετικά συζητήσεις, υπάρχουν πολλοί ειδικοί για αυτό το θέμα, αλλά νομίζω και εδώ δεν θα πρέπει να ονειροπολούμε. Ε, ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις. Δηλαδή η, η μετανάστευση μπορεί να αμβλύνει τα δημογραφικά προβλήματα αλλά δεν μπορεί να αλλάξει ριζικά το, τοπίο, της το δημογραφικό τοπίο. Γιατί υπάρχουν χώρες που γυράσκουν και εντός του ΩΣΑ. Επίσης υπάρχουν κάποια όρια στις ε, προοπτικές ανοίγματο μετανάστευσης που έχουν σαν αποτέλεσμα έστω και αν κρατάμε το επίπεδο των ε, ρευμάτων εισρωής που είναι ιδιαίτερως υψηλό τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, έστω και τότε δεν θα, δεν θα μπορούσαμε να ρυθμίσουμε το πρόβλημα της απασχόλησης και ανάπτυξης σε ορισμένες χώρες που είναι χώρες μετανάστευσης και που θέλουν να είναι ακόμα περισσότερο χώρες μετανάστευσης. Λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές εδώ και να οριοθετήσουμε σωστά το πρόβλημα και να μην ε, στηριζόμαστε υπερβολικά στην ε, μετανάστευση. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μείωση των εμβασμάτων σήμερα. Νομίζω ότι πρόκειται μια, ε, διαμάχη, μια μάχη μάλλον ε, στην οποία θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τα όπλα μας γιατί δεν θα πρέπει τα εμβάσματα να υποκαθιστούν τον όγκο βοήθειας που θα πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνονται και όχι να υποκαθίστανται από άλλες μορφές ε, μεταφορών κονδυλίων που σε περίοδους κρίσης είναι ιδιαίτερως αβέβαιες. Δεν έχουμε πολύ χρόνο γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και πρέπει και εσείς να πάρετε το λόγο και να θέσετε ερωτήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να αφιερώσω το λίγο χρόνο που μου απομένει σε δύο θέματα. Δηλαδή να δούμε τι γίνεται με την ε, μετανάστευση της εργασίας στις χώρες του ΩΣΑ είτε μπορεί να προωθηθεί από τους εργοδότες τροποτινά και αυτό υφίσταται. Σήμερα το πρωί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, μια ενδιαφέροντα, ενδιαφέρουσα ομιλία μάλλον εκ μέρους του εκπροσώπου των μεγάλων πολυεθνικών ο οποίος μιλάει για ένα τεράστιο άνοιγμα στην αγορά της εργασίας. Ε, ξέρουμε ότι σήμερα ε, ε, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υποφέρουν περισσότερο. Γι' αυτό υπάρχει πολύ παράνομη εργασία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όχι επειδή προτιμούν οι εργοδότες τους παράνομους, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσλάβει κανείς έναν αλλοδαπό, ε, εκτός αν είναι βεβαίως προέρχεται μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεχομένω λοιπόν κάποιες διαδικασίες προωθούνται από τους εργοδότες. Αλλά όταν υπάρχει ανεργία ε, δεν υπάρχει μετανάστευση. Άλλες διαδικασίες, δεύτερος τύπος ε, διαδικασιών, αυτές προσωμιάζουν στις διαδικασίες του Καναδά ή των Ηνωμένων Πολιτειών, Γερμανίας, Γαλλίας κλπ. όπου είναι η χώρα αυτή η οποία ασκεί τον έλεγχο, διαχειρίζεται την μετανάστευση. Κάτι το οποίο δεν είναι κατά ανάγκη αρνητικό, γιατί η οποια ασκει τον ελεγχο διαχειριζεται την μεταναστευση κατι το οποιο δεν ειναι κατα αρνητικο γιατι η ιστορια της μετανάστευσης είναι και ιστορία ε, των ε, ιδιωτών οι οποίοι παρέχουν ενδιάμεσον που προσφέρουν εργατική δύναμη κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι πολύ ρόδινα ούτε από την πλευρά των εργοδοτών ούτε από την πλευρά των χωρών. Όταν θέλουμε να θέσουμε τη συζήτηση αυτή, η μετανάστευση, η ανάπτυξη, θα πρέπει να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τι χώρε προέλευση και αυτό δεν είναι πάντοτε προφανές ή πολύ απλό να επιτευχθεί. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, δηλαδή η παράνομη μετανάστευση, ε, η παράνομη απασχόληση αλλοδαπών, ε, το γεγονό ότι υπάρχουν τεράστια ποσοστά ανεργία μεταξύ μεταναστών. Τα παιδιά των μεταναστών που έχουν εκπαιδευτεί στι χώρε υποδοχή δεν μπορούν να βρουν εργασία και ακόμα και όταν είναι, έχουν υψηλό επίπεδο εξειδίκευση, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά παράδοξο. Δηλαδή, ε, οι χώρες που θέλουν εξειδικευμένο δυναμικό είναι γεμάτες από ανθρώπους που έχουν υψηλά προσόντα, είναι ιδιαίτερως ειδικευμένοι και τελικά καταλήγουν όμως να κάνουν δουλειές χαμηλής ειδίκευσης ή ανειδίκευτες. Θα ήθελα να ε, θέσω τώρα τέσσερα ερωτήματα για να τα βάλω εδώ στο τραπέζι ε, της συζήτησης. Ε, το πρώτο είναι, αναφέρθηκε άλλωστε σήμερα το πρωί, κατά πόσο τι γίνεται με την προσωρινή μετανάστευση. Υπάρχουν κάποιες θέσεις εργασίας των οποίο έχουμε ανάγκη και που δεν θέλει κανείς να τις καλύψει, έστω και σε περίοδος κρίση. Ε, το να μαζεύει κανείς τα σκουπίδια ή σε κάποιους κλάδους που είναι εξαιρετικά ανεπιθύμητοι. Ε, ο δεύτερος, ε, το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να θέσω είναι το τι πρέπει να γίνει για να αναπροσανατολίσουμε την παράνομη μετανάστευση σε κανονικού νόμιμους διάβλους. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Σε χώρε όπω είναι η Ισπανία, εγώ προσωπικά ε, εμένα προσωπικά μου άρεσε πολύ η παρέμβαση τη κυρίας Μπλάνκο, γιατί η Ισπανία είναι μια χώρα η οποία υποδέχθηκε εκατομμύρια μεταναστών. Ε, είναι 10 ή 12 εκατομμύρια είναι μια χώρα η οποία ανέπτυξε μια εξαιρετικά πρωτότυπη πολιτική μετανάστευσης και πραγματικά ήταν υποδειγματική στους κόλπους του ΩΣΑ. Αλλά το μοντέλο αυτό ε, κατέρευσε ή μάλλον δέχτηκε πολλές επιθέσεις από τα μέσα μαζικής ε, ενημέρωσης γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που προσπάθησαν να πάνε στην Ισπανία ε, για να κερδίσουν το ψωμί τους πέθαναν και όλη η πολιτική της Ισπανίας τελικά καταστράφηκε από αυτές τις συμπεριφορές που κατέστησε εξαιρετικά δυσχερή τη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών. Αυτό το θέμα συνδέεται επίσης με την συνεκτική πολιτική ανάπτυξη. Ε, τρίτον, τι μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο αυτό που είναι ακριβώς η οικονομική συγκυρία της κρίσης. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην... Ε, ε, ε, ε, να μην εγκαταλείψουμε ε, τους μετανάστες να προσπαθήσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική, να κάνουμε τα πάντα ούτως ώστε τα παιδιά των μεταναστών να εκπαιδεύονται σωστά να μπορούν να βρουν μια εργασία. Δεν θα πρέπει να περιζόμαστε στο, στην προβληματική των εμβασμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να χαράξουμε μια σωστή ολοκληρωμένη πολιτική χωρίς να επιτρέπουμε τελικά να εκτροχιάζεται η, η σκέψη μας ε, προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Τώρα, πώ μπορούμε να βελτιώσουμε την πολιτική ανάπτυξη. Νομίζω θα πρέπει καταρχήν να μειώσουμε τα εμπόδια στην κινητικότητα τη εργασία, κάτι το οποίο προτάθηκε προηγουμένω και αυτό μπορεί να γίνει με έναν δημαγωγικό τρόπο, λέγοντα ότι πρέπει να κάνουμε τεράστιο άνοιγμα κλπ. ή μπορούμε να το κάνουμε πιο ισορροπημένα, προτείνοντα μια μορφή συνεργασία, ώστε η κανονική νόμιμη μετανάστευση να έχει την ε, πρωτοκαθεδρία. Δηλαδή, όσον αφορά την ε, ε, τα εμβάσματα, είναι σκανδαλώδες οι προμήθειες της τάξης του 20%. Ε, θα πρέπει να έχουμε το κουράγιο να πούμε ότι σε πολλές χώρες προέλευσης τα ε, συστήματα αυτά των συναλλαγών πραγματικά είναι απαράδεκτα και γίνονται προσπάθειες σήμερα με τις νέες τεχνολογίες να καταργηθούν αυτές οι σκανδαλώδεις αστρονομικές προμήθειες μέσω των νέων τεχνολογιών. Τώρα, όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση των μεταναστών, δεν είναι πρόβλημα να έχουμε εξειδικευμένους μετανάστες. Το θέμα είναι να ξέρουμε ποιος πλήρωσε για την εκπαίδευσή τους και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε μορφές συνεργασίας και βοήθειας, ούτως ώστε εάν ε, εκπαιδευτούν 100 νοσοκόμε στη Ρουμανία και πάνε 20 στην Ευρώπη, τουλάχιστον 80 να μείνουν στη χώρα του. Πώ ε, πώς μπορεί να γίνει μια αποκέντρωση επίση σε χώρε όπω η Ιταλία κλπ. Θα πρέπει να αναπτυχθούν τέτοιε μορφέ συνεργασία. Νομίζω έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου και επίση έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να κλείσω την ομιλία μου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκαρσόν. Ευχαριστώ τους και τους δύο μιλητές και τώρα ε, ασχολούμεθα με το πρώτο πάνελ που έχει τίτλο με το κύριο θέμα του πάνελ έχει τίτλο μετανάστευση και ανάπτυξη από την ε, κοπτική γωνία των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Ο κύριος Ντέιτον είναι από τον ΩΣΑ. Ε, ο κύριος Ντάμπη, ο κύριος Μαυρομάτης, Μπάση Ρουντιάρα και Τζον Πάτελ παρακαλώ να έρθουν εδώ. Δίνω το λόγο κατευθείαν στον κύριο Ντέιτον Τζόνσον και τον παρακαλώ να μην ξεπεράσει τα 30 λεπτά. Euh, και για να υπάρχει και χρόνος μετά για ερώτα απαντήσεις. Καλησπέρα σας. Έχουμε μαζί μας πολλούς και γνωστούς ε, ομιλητές προτείνω να ακολουθήσουμε, είμαστε πειθαρχημένοι να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα όπως θα δόθηκε ξεκινούμε από τον κύριο Ντάμπι που είναι από την Αυστραλία βουλευτής ασχολείται με θέματα ε, εξωτερικής πολιτικής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. και ο οποίος είναι και στην Διοικητική Επιτροπή του Παγκόσμιου Κινήματος ε, στη Washington. Ντάμπι, ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε εδώ. Ελπίζω η προφορά μου από την Αυστραλία να μην με κάνει δυσνόητο από τον, παγκόσμιο, από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πάνω από 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι ε, μετανάστευσαν στην Αυστραλία σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό των 21 εκατομμυρίων ε, αναλογικά δηλαδή η Αυστραλία είναι μεγαλύτερος υποδοχέας ε, μεταναστών η ξένοι μετανάστες στην Αυστραλία παίζουν τεράστιο ρόλο ε, σε όλους τους τομείς και πιστεύουμε ότι μας βελτίωσαν. Η, κατά κύριο λόγο υπήρξαν κέρδη από την μετανάστευση στη χώρα μου για και στα οικονομικά και στο, ε, στις κοινωνικές εκδηλώσεις, στα παιδιά μας, στον αθλητισμό. Ε, μας κάνανε μια κοσμοπολίτικη κοινωνία τελικά. Και τα δύο είναι οι βασικοί πυλώνες που ε, εφαρμόζουμε στην πολιτική μας πρώτον αυτόματα ο μετανάστης μετά από δύο χρόνια παραμονής στη χώρα μας γίνεται παίρνει την α, ε, υπηκότητα τη δική μας και δεύτερον ε, δεύτερο βασικός πυλώνας είναι ο σεβασμός και η τήρηση αν θέλετε βασικών αρχών δημοκρατικού ήθους κτλ. Επίσης τώρα για όσον αφορά τη μετανάστευση υποστηρίζουμε τη μόνιμη μετανάστευση αν θέλετε αυτούς που έρχονται στην Αυστραλία για να μείνουν και βεβαίω οι, οι Αυστραλοί δεν ήταν πάντα υπέρ των μεταναστών πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν κατά όταν ο δικός μου πατέρας έφτασε στην Αυστραλία το 1939 σαν Γερμανός μετανάστη μετανάστη από τη Γερμανία θεώρησε ότι οι ντόπιοι ήταν κυρίως ήταν τελείως εχθρικοί και ακόμη πιο εχθρικοί απέναντι στους Γερμανούς το Τη δεκαετία του 30 του 40 η Αυστραλία δέχτηκε πάρα πολλούς μετανάστες από όλη την Ευρώπη ε, Τουρκία και Λουιβανός ε, μας, μας έστειλαν μετανάστες ε, το 60 και τώρα έχουμε μετανάστες και από την Καμπότζη ε, πριν από την ε, χρηματοπιστωτική κρίση ε, δεχτήκαμε γύρω στους 200.000 μετανάστες ε, και μάλιστα με προσόντα και ικανότητες και αυτοί βοήθησαν οικονομικά την Αυστραλία ιδιαίτερα όταν δεν είχαμε το εργατικό δυναμικό με τα προσόντα που ε, απαιτούσαν, απαιτούσαν οι θέσεις εργασίας και η χώρα μας ανέκαθεν πιστεύει ότι η μετανάστευση είναι κομμάτι όλων των πολιτικών και επιδιώκουμε συνοχή στις πολιτικές μας. Βεβαίως οι Άγγλοι και οι Ζηλανδοί είναι οι κύριοι μετανάστες. Ε, από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι από την Νότια Αφρική και από... Ε, άλλες αγγλόφωνες χώρες ε, τα τελευταία χρόνια όμως βλέπουμε και λάθρο μετανάστευση ιδιαίτερα από την Ασία και Ανατολική Ασία και Μέση Ανατολή που ε, ζητούν ε, ε, να γίνουν πρόσφυγες έρχονται ως πρόσφυγες στην Αυστραλία στην πρόσφατη επίσκεψή μου ε, στο Γερμανία έμαθα ότι 350.000 ήταν οι μετανάστες το 2000 στη Γερμανία ενώ σε εμάς ήταν 400.000 πιστεύουμε ε, ότι όπως σας είπα αναλογικά έχουμε πάρα πολλούς μετανάστες σε σχέση με τον τόπιο πληθυσμό ε, εμείς πιστεύουμε βέβαια ότι η είσοδος των μεταναστών αυτών θα πρέπει να γίνει με τακτικό τρόπο βεβαίως έχουμε και προβλήματα όπως με τους boat people από την Ινδονησία με αυτούς που έρχονται με τα καραβάκια από την ε, Ινδονησία και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα γιατί, αλλά βέβαια το πρόβλημα είναι κατανοητό γιατί η Ινδονησία είναι κοντά στην Αυστραλία τελικά. Τώρα από εκεί και πέρα ο κύριος Αμάνου μίλησε και για ε, ε, κάποιους που χρησιμοποιούν τελικά λαϊκιστικές προσεγγίσεις γιατί αυτό αρέσει στον κόσμο και με αυτή την έννοια υποδαβλίζουν και ξενοφοβία και τα Όχι, εμείς προσπαθούμε να μην κάνουμε κάτι τέτοιο. Πιστεύουμε ότι αυτού του είδους προσέγγιση είναι λάθος και για τη διαρροή εγκεφάλων το brain drain που ετέθη από τον κύριο Γκαρσόν πριν από λίγο εμείς ε, ένα σε εμά ένα εκατομμύριο από, τους, από τα 21 εκατομμύρια κατοίκους μας είναι ξένοι αν θέλετε είναι μετανάστευση ε, ε, είναι μετανάστες αλλά σε μόνιμη βάση ε, πιστεύουμε ότι επίσης ότι και προσπαθούμε να κάνουμε ε, πολλά πράγματα για τους μετανάστες και για τη μετανάστευση κάνουμε, οργανώνουμε εκδηλώσεις, συνέδρια ε, φαρμό, ε, δίνουμε το λόγο στους μετανάστες σε αυτούς που έρχονται πρόσφατα όπως σας είπα ως πρόσφυγες έχουμε έναν διαμεσολαβητή για, το, για θέματα μετανάστευσης και υπάρχει Υπουργείο Μετανάστευσης ε, και κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι παρά την οικονομική κρίση τώρα και τα, τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές στην Αυστραλία πιστεύουμε ότι η μετανάστευση μπορεί βέβαια να μειωθεί λιγάκι αλλά δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Μπορεί απλώς να γίνει λίγο μικρότερη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Μανώλης Μαυρομάτης από την Ελλάδα που εξελέγει Ευρωβουλευτής το 2004. Είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής για Μετανάστευση Πολιτισμό κτλ. Και, ε, και έχει και πολλά άλλα καθή... καθήκοντα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί και αγαπητέ συνάδελφοι, φίλοι προσκεκλημένοι, είναι γεγονός ότι υπάρχουν στον κόσμο 175 εκατομμύρια μετανάστες αριθμός που σχεδόν τριπλασιάστηκε τα τελευταία 40 χρόνια. Δεν πρόκειται όμως ε, για ένα νέο φαινόμενο. Οι διαστάσεις που έχει λάβει η μετανάστευση στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της πρόσφατης οικονομικής κρίσης μας φέρνει καθημερινά αντιμέτωπους με ανθρώπινες τραγωδίες. Η φτώχεια, η ανέχεια, η απόγνωση, η στέρηση βασικών ελευθεριών και δικαιωμάτων οδηγούν χιλιάδες Αφρικανούς στις βόρειες ακτές της Μεσογείου ή στα Κανάρια νησιά και εκατοντάδες ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η μόνη αντίδραση των ευρωπαϊκών κρατών συνίσταται στην αύξηση των ελέγχων και των περιπόλων που αναγκάζουν τους ανθρώπους να διατρέχουν ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους στην ε, προσπάθειά τους να έρθουν στην Ευρώπη. Τα σύνορα όμως της Ευρώπης δεν είναι αδιαπέραστα. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα μέσα που ήδη υπάρχουν. Κυρίως όμως οφείλουμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας. Βέβαια η αύξηση της βοήθειας δεν αποτελεί από μόνη της τη λύση. Η δημοσιονομική ενίσχυση είναι ένα από τα ανεγνωρισμένα μέσα αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω από το 20% των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης δαπανώνται ήδη για το σκοπό αυτό και η τάση είναι αυξητική. Αν υπάρχει το σωστό πλαίσιο, η δημοσιονομική ενίσχυση μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας. Οι χορηγοί και οι αποδέκτες επιλέγουν μια εταιρική προσέγγιση στην αναπτυξιακή συνεργασία η συμφωνία για την ενίσχυση αναπτυξιακών στρατηγικών και προγραμμάτων του αποδέκτη και κυρίως για εκτενείς στρατηγικές για την καταπολέμηση της στόχιας αποτελεί βασική προϋπόθεση της συμφωνίας αυτής. Το ζητούμενο δεν πρέπει να είναι μόνο η εκταμείευση των πόρων ή η διαβεβαίωση της σωστής χρησιμοποίησής τους. Θα πρέπει πάντα να εξετάζεται και η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής ενίσχυσης από τη σκοπιά του αν επιτυγχάνονται καλύτερα οι επιδιωκόμενοι στόχοι μέσω της χρηματικής βοήθειας παρά με άλλα οποιαδήποτε μέσα. Παρ' όλα αυτά όλοι συμφωνούμε πιστεύω ότι η δημοσιονομική βοήθεια δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν δεν είναι διαφανής, υπεύθυνη και αποτελεσματική η διαχείριση των δημοσίων δαπανών από την πλευρά του αποδέκτη. Γνώμη μου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να λάβει μέτρα στα μέρη όπου βρίσκονται οι μετανάστες, στα μέρη από όπου ξεκινάει η μετανάστευση. Είναι εύκολο να προσδιοριστούν οι κύριες περιοχές μετανάστευσης, εφόσον πρόκειται συνήθως για τις φτωχότερες και να χρηματοδοτηθεί βεβαίω η δημιουργία υποδομών προκειμένου οι άποροι πληθυσμοί να έχουν λόγους παραμονής. Δρόμοι, κέντρα υγείας, σχολεία, πόσιμο νερό, αηφόρος καλλιέργεια. Η χρηματοδότηση βοήθειας σε ιατροφαρμακευτικό υλικό ή τρόφιμα δεν λύνει ασφαλώς το πρόβλημα. Η ουσία είναι να βοηθήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάπτυξη υποδομών που σταδιακά θα βγάλει τους κατοίκους των περιοχών αυτών από την ανέχεια, θα τους παρέχει αυτονομία, εξέλιξη και ως εκ τούτου θα περιορίσει την κινητικότητά τους. Είναι εξίσου εύκολο να προσδιοριστούν οι μεταναστευτικοί πόλοι Πρόκειται για τα κράτη ή τις μεγάλες πόλεις που διαθέτουν σύγχρονα μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας και που αποτελούν εξίσου σημεία υποδοχής και αναχώρησης για τις μεγάλες οδούς μετανάστευσης. Με τον προσδιορισμό των πόλων και των πηγών μετανάστευσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση να εφαρμόσει ακόμα περισσότερες δράσεις από τις σημερινές, πιο αποτελεσματικές που θα έχουν στόχο κυρίως την ενίσχυση των πληθυσμών και επιπλέον των πιο ευάλωτων ομάδων όπως οι γυναίκες και τα παιδιά. Τέλος, θα μπορούσε να καθιερωθεί ένα πρόγραμμα ενημέρωσης γιατί αυτές οι ζώνες είναι οι πλέον ευάλωτες. Και αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης θα προορίζεται και θα προορίζεται αποκλειστικά για μετανάστες. Όσον αφορά τώρα την ενσωμάτωση, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει την αξιοποίηση του δυναμικού που παρουσιάζουν οι κοινότητες των μεταναστών που έχουν συγκροτηθεί ήδη μετά την μετανάστευση. Θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση που θα μετατρέψει τους μετανάστες σε πρωταγωνιστές της ανάπτυξης στο όνομα της συνοχής και της αλληλοβοήθειας. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να προωθήσουμε τις μεταφορές κονδυλίων στις χώρες προέλευσης να τα καταστήσουμε πιο διαφανή, λιγότερο δαπανηρά και να μελετήσουμε ένα νέο οικονομικό προϊόν που θα μπορούσε να λάβει τη μορφή ενός σχεδίου αναπτυξιακής αποταμίευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της πρέπει να εφαρμόσουν καινοτόμες πολιτικές όπως η ανάληψη ευθύνης για την επιστροφή των μεταναστών που το επιθυμούν βεβαίως στη χώρα προέλευσή τους κυρίως τους ερευνητές και τους γιατρούς στο πλαίσιο θεσμικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και νοσοκομείων. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε την κυκλική μετανάστευση, επιτρέποντας στους μετανάστες να αναχωρούν και να επιστρέφουν σε συνεργασία ασφαλώς με τις χώρες προέλευσης και διασφαλίζοντας τη μεταφορά κοινωνικών παροχών. Ένα τέτοιο μέτρο κατά την προσωπική μου γνώμη θα εξάλληφε σταδιακά την διαρροή των λεγόμενων εγκεφάλων και θα επέτρεψε και θα επέτρεπε την κυκλοφορία των πραγματικών εγκεφάλων. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες η μετανάστευση είναι συνώνυμη της αποδημίας των ατόμων με την καλύτερη μόρφωση ή το εντονότερο επιχειρηματικό πνεύμα αυτό έχει δραματικές επιπτώσεις για τις φτωχές αυτές χώρες από τη στιγμή που το φαινόμενο επηρεάζει συχνά βασικούς τομείς όπως η υγεία, η έρευνα και η εκπαίδευση. Τα θέματα τα οποία σας ανέπτυξα είναι στην εισήγησή μου ως γνωμοδότης για την νόμιμη και παράνομη μετανάστευση στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ για την ε, παρέμβαση και γιατί τε, παραμείνατε μέσα στα χρονικά όρια. Ο επόμενος ομιλητή είναι ο κύριος Μπασιρού Ντιάρα που είναι σύμβουλος του Πρόεδρου του Μαλή. Ο κύριος, κύριε Ντερά, έχετε το λόγο. Je vous euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να παρέμβω εδώ στην Ομίγυρη σχετικά με θέματα μετανάστευσης και πιο συγκεκριμένα για το θέμα της συνεκτικότητας των πολιτικών που πρέπει να υπάρχει Εγώ θα ασχοληθώ λίγο παραπάνω με το θέμα της συνανάπτυξης και της ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων και θα πω και μερικά λόγια για το κέντρο που ε, ιδρύθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 2008 στη χώρα μου. Ε, όταν μιλάω για συνανάπτυξη θα αναφερθώ προφανώ στη συνεργασία Γαλλίας-Μαλή. Το 98 το το 1998 έγιναν συζητήσεις και σοβαρές ε, αναλύσεις μεταξύ δύο χωρών για το φαινόμενο της μετανάστευσης μεταξύ Γαλλίας και Μαλή και στις 14 Μαρτίου του 2001 μια επιτροπή γαλλο-μαλική και εγώ ήμουν πρόεδρος εκείνης της Επιτροπής εκ μέρους του Μαλή ε, μια τέτοια επιτροπή λοιπόν και τέσσερις τεχνικές επιτροπές συστάθηκαν για να ασχοληθούν με όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση. Η πρώτη τεχνική επιτροπή ε, που συστάθηκε είναι η Επιτροπή της του co-development όπως λέμε αυτής της συνανάπτυξης ε, δεν υπάρχει επιτροπή που ασχολείται με την κυκλοφορία μεταξύ των δύο χωρών θεωρήσεις, διαβατήρια κλπ μετά υπάρχει μια τεχνική επιτροπή για που συζητεί θέματα ε, στέγασης ε, παιδιών δεύτερης τρίτης γενιάς ε, επασχόλησης, οικογενειακή ζωή κτλ. Και τελικά υπάρχει μια τέταρτη τεχνική επιτροπή που ασχολείται αποκλειστικά με θέματα νεότητας νέων αυτοί, αυτές λοιπόν οι επιτροπές είναι η βασική δόμη που φτιάξαμε για να μπορέσουμε να συζητήσουμε ε, τη συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Μαλή για θέματα μετανάστευσης και ανάπτυξης. Η Επιτροπή, όπως σας είπα ήμουν εγώ ε, στην Επιτροπή της Συνανάπτυξη η οποία υπέβαλε την έκθεσή της στη Γερουσία ε, στη Γαλλία μετά από λίγο χρόνο, από ε, λίγο καιρό και η οποία συνεχίζει βεβαίως τις εργασίες της γιατί υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία αλλιώς τα βλέπει η Γαλλία, αλλιώς τα βλέπουμε εμείς. Αυτά τα θέματα πρώτα-πρώτα λοιπόν πρέπει να ξεκαθαριστούν και πρώτα-πρώτα η έννοια του co-development. Τι είναι η συναπτά, συνανάπτυξη. Είναι ένα εργαλείο στην περίπτωση μιας εταιρικής σχέσης που εξυπηρετεί τη χώρα προέλευσης το ουσιαστικά το μετανάστη προσπαθεί να τα αξιοποιήσει τα θετικά που υπάρχουν και επίσης είναι και ένα εργαλείο διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών <clears throat> και ασχολείται αν θέλετε, περιλαμβάνει και την επιστροφή στη χώρα προέλευσης του μετανάστη η πολιτική τώρα της ενανάπτυξης και το περιεχόμενό της αλλάζουν αυτά βέβαια ανάλογα με τη χώρα περί της οποίας πρόκειται Μαρόκο, Γαλλία η Μαλή, Γαλλία δεν είναι το ίδιο πράγμα οι διαφορές ε, ερμηνείας ουσιαστικά που υπάρχουν ε, επηρεάζουν φυσικά και τα αποτελέσματα που τα οποία προσδοκά κανείς από την πολιτική συνανάπτυξη. Η Γαλλία και το Μαλί ήταν οι πρόδρομες χώρες της συνανάπτυξης πρέπει να πω και δεν μπορούμε αυτή τη συνανάπτυξη να τη δούμε ξεχωριστά από από δράσεις που ανελήφθησαν υπέρ των μεταναστών που, του μεταναστευτικού κύματος της δεκαετίας του 60 γιατί υπήρχαν επιτυχίες σε σχέση με αυτούς τους μετανάστε. μετανάστες επίσης δεν πρέπει να, τα, αγνοήσουμε αυτά που έχουν γίνει και σε κοινοτικό επίπεδο κατάρτιση, επιμόρφωση, πρόσβες στο πόσιμο είδος, είδωρ κλπ. Στην ε, Γαλλία υπάρχουν 400 σύλλογοι περίπου ε, υπηκών του Μαλή οι οποίοι στο καταστατικό τους έχουν βάλει και την ιδέα, τις ιδέες και οι αξίες αυτές της συνανάπτυξης θέλουμε η συνανάπτυξη να γίνει σημαντικός μοχλός ανάπτυξης και της μετανάστευσης και των χωρών ε, από τους οποίους προέρχονται οι μετανάστες. Θέλουμε οι μετανάστες να είναι πραγματικοί φορείς ε, ενεργοί στην ανάπτυξη μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και της χώρας υποδοχής, χώρας προορισμού και της χώρας προέλευσης. Ξε, επίσης φτιάχτηκε μια διυπουργική αποστολή στο Μαλί για το θέμα της συνανάπτυξης και ε, η πολιτική συναναπτυξη κατέληξε στις 21 ε, Μαΐου του 2000 στην υπογραφή μιας σύμβασης με επίσημες με το Μαλή ε, η τελική συμφωνία μετά τις επικυρώσεις έγινε το 2002 και μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια ε, τα σχετικά κονδύλια για την πρώτη φάση. Η σύμβαση αυτή τι περιλαμβάνει. Περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια ουσιαστικά. Πέντε συνιστώσεις ε, για την ανάπτυξη των ε, γενική ανάπτυξη, τοπική ανάπτυξη, ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εμπορικών επιχειρήσεων, ε, νεότητας, μετανάστευση κτλ. Και η πέμπτη συνιστόσα ε, είναι η διαχείριση των διαφόρων σχεδίων. Στις 15 Μαρτίου του 2006 υπεγράφει η σύμβαση για τη δεύτερη φάση. Άλλα τρία χρόνια πάλι 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η δεύτερη φάση ε, εκπνέει ε, όπου να είναι και ε, θα δούμε πώς θα συνεχιστεί η υπόθεση αυτή. Μπορούμε, φαντάζομαι, να φανταστούμε όλοι μας ότι καλό θα ήταν να γίνει ένας απολογισμός της πολιτικής συνανάπτυξης και ίσως θα έπρεπε να έχει γίνει 7-8 χρόνια αργότερα εγώ εκείνο που λέω είναι το εξής ότι ακόμη δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτά που είχαμε θέσει σαν στόχους. Δεν μπορέσαμε να αναπτύξουμε στο εσωτερικό της, να, να να κάνουμε πράγματα που θα βοηθούσαν η, τη μετανάστευση να αποδειχθεί βασικός πυλώνας ανάπτυξης και της χώρας προέλευσης. παρόλα όλα αυτά υπήρχαν διάφορα προγράμματα ε, πολλά σχέδια, 22 σχέδια σε επίπεδο τοπικής αυτοδίκης, 300 περίπου σχέδια ε, ε, α, σε χαμηλότερο επίπεδο εκατοντάδες σχέδια ε, υπήρχαν κατά 63% η χρηματοδότηση αυτών των ε, σχεδίων έγιναν από δημόσια κονδύλια 29 από τους ίδιους τους μετανάστες και 8% από άλλες ιδιωτικές πηγές Τώρα, ε, άλλα πράγματα, οι ε, επενδύσεις εξ αποστάσεως που συζητάγαμε, τα βιβλιάρια αν θέλετε από τα ε, που συζητούσαμε στην αρχή παρέμειναν όνειρο δεν υλοποιήθηκαν ποτέ εδώ που βρισκόμαστε λοιπόν το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπολείπονται πολύ τα επιτεύγματα από τις προσδοκίες που υπήρχαν και γι' αυτό αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να βοηθήσει να βοηθήσει στο να διευκρινιστούν ορισμένες βασικές έννοιες του co-development όπως το ονομάζουμε και να προωθηθεί περαιτέρω η ιδέα αυτή η συνανάπτυξη αυτή και να οδηγήσει τον μετανάστη σε πιο παραγωγικούς τομείς να σχετιστεί με την απασχόληση και τη θέση εργασίας που θα βρει ο μετανάστης κτλ. Να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα για το κέντρο ενημέρωσης και κατάρτιση των μεταναστών ο Επιτρόπος Λουί Μισελ ε, στις 6 Οκτωβρίου στον Παμάκο ε, το κέντρο αυτό το, το οποίο η έμπνευση προέρχεται από την ε, ε σύμβαση του Ραμπά και της Τρίπολης μετά το 2006 και το κέντρο αυτό θα ήταν ένα κέντρο πιλότος θα γινόταν και άλλα τέτοιου είδους κέντρα στην Δυτική Αφρική της 23 Οκτωβρίου του 2007 υπεγράφει η Συμφωνία για τη Χρηματοδότηση και ε, ορίστηκαν και οι στόχοι ε, του κέντρου αυτού το οποίο έχει σαν στόχο να φτιάξει, ένα στόχος του είναι να φτιάξει μια βάση δεδομένων για την μετανάστευση στην περιοχή ε, μια βάση δεδομένων για τους μετανάστες που επιστρέφουν στις χώρες προέλευσης μια, μια βάση δεδομένου για τους λαθρομετανάστες και για μέτρα πρόληψης της λαθρομετανάστευσης και πείστε υπάρχουν και άλλοι στόχοι βεβαίως του κέντρου αλλά εκείνο που πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνει το κέντρο αυτό είναι να συνεργάζεται και με άλλες διοικητικές αρχές παραδείγματο χάρη με το Υπουργείο Απασχόλησης με μη κυβερνητικέ οργανώσεις κτλ. Και ε, ε, ε Πραγματικά ε, το κέντρο αυτό άρχισε να λειτουργεί αλλά το, δεν λειτουργεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορούμε να κάνουμε αξιολόγηση. Ευχαριστώ. Ο τελικός ομιλητής αυτού του πάνελ είναι ο κύριος Τζον Μπάτλ που είναι ε, βουλευτής στο Λίτς, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν ε, υπουργός εξωτερικών πολλές φορές ασχολείται με θέματα ανάπτυξης, τον απασχολούν πάρα πολύ. Επίσης είμαι εκπρόσωπος ε, στο Global Action. Ευχαριστώ. Παρότι είμαι μέλος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που παρακολουθεί τις Υπουργές του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν την ανάπτυξη και την ε, ε, βοήθεια, νομίζω ότι θα έπρεπε να τονίσω ότι δεν θα ήμουν στο Κοινοβούλιο αν δεν με είχε εκλέξει η γειτονιά μου. Και θα ήθελα να δώσω έτσι και ένα πολιτικό ρεαλισμό σε αυτή τη συζήτηση τη σημερινή. Η γειτονιά μου είναι ε, μια κλασική περίπτωση έτσι υποβαθμισμένης γειτονιάς. Ε, αποτελείται από ημικαταρτισμένους ε, εργαζομένους ε, και όταν η οικονομία ε, είναι σε ύφεση είναι οι πρώτοι που χάνουν τη δουλειά τους από το 7% ε, φτάσαν στο 12% ε, το 2008 ε, σε σχέση με το 2000 οι μετανάστες. Και πολύ κοντά στο σπίτι μου μιλούνται 26 γλώσσες. Η πόλη μου χτίστηκε από Ιρλανδούς εργάτες που ήταν μετανάστες στο Λίτζ. Δεν θα ήμασταν εδώ που ήμασταν στο Λίτζ δηλαδή, αν δεν είχαν έρθει οι Ιρλανδοί, αν δεν είχαν έρθει οι Ινδοί και τα λοιπά να δουλέψουν στα κλωστεφαντουργία κτλ. Ε, να δουλέψουν στις μεταφορές και πρέπει να τονίσω ότι σήμερα στην εκλογική μου περιφέρεια εάν φεύγαν οι μετανάστες θα είχαμε τεράστια προβλήματα για να φροντίσουμε τους ε, ηλικιωμένους. Υπάρχουν λοιπόν και αν φεύγανε θα είχαμε τεράστια προβλήματα. Λοιπόν, γιατί αναφέρω την ε, εκλογική μου περιφέρεια και την γειτονιά μου. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η συνοχή στην αναπτυξιακή πολιτική, σε τοπικό, σε εθνικό ή σε διεθνέ επίπεδο. Η δική μου εκλογική περιφέρεια θα ήθελε να υπάρχει τέτοια συνοχή, γιατί έχει συχαθεί αυτές τις αντιφάσεις ε, που υπάρχουν στις πολιτικές μας. Πρέπει να πείσω τους ε, εκλογείς μου, και συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλια που ακούστηκαν, ότι εμείς στη Βρετανία θα πρέπει να συνεχίσουμε την ε, αναπτυξιακή μας βοήθεια και να κρατήσουμε αυτή την γραμμή στο προπολογισμό. Πρέπει να επιστρέψω στους εκλογείς μου και να τους εξηγήσω γιατί ένα τμήμα από τους φόρους που πληρώνουν πρέπει να πάει στην αναπτυξιακή βοήθεια. Κάτι που, πάει καλά, που, κάν, που κάναμε καλά στην Επιτροπή μου είναι αυτό το κείμενο πώς η μετανάστευση θα βοηθήσει στη μείωση της στόχης. Αυτό το δημοσίευσαμε το 2003. Τις τελευταίες εβδομάδες, στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης, ε, φτάσαμε και μιλήσαμε με τους ε, υπουργούς και με τα άλλα κόμματα για να τους πείσουμε ότι θα πρέπει η αναπτυξιακή βοήθεια να είναι η ε, ιερή και απαραβίαστη, να μην τη μειώσουμε λόγω της κρίσης. Και συμφωνήσαμε. Και είναι σημαντικό αυτό που συμφωνήσαμε. Τώρα πάω στο θέμα της μετανάστευσης θα πρέπει να θεωρήσουμε ε, ότι η μετανάστευση ε, είναι επωφελής και για τους μεν και για τους δε. Και θέλω να μιλήσω για την, την έννοια της συνανάπτυξης ε, που είπατε εσείς. θα μπορούσα να σας δώσω αριθμητικά στοιχεία για το πόσο κερδίζουμε οικονομικά ε, εμείς. μας δίνουν 6 δισεκατομμύρια το χρόνο. Αν φεύγανε η οικονομία μας θα συρρυκνωνόταν. Ακόμα και σήμερα με την οικονομική κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε θετικοί για την ε, μετανάστευση. Χρειάζομαι όμως την υποστήριξη των εκλογέων μου. Και η πρόκληση είναι η εξή. Μέσα στα πλαίσια της παγκόσμιας κρίσης θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η μετανάστευση δεν είναι νέο φαινόμενο, δεν είναι αποκατάσταση της ε, ανάπτυξης, δεν είναι υποκατάστατο η αποτυχία της ανάπτυξης. Υπάρχει. Και υπάρχουν, ε, υπάρχει μετανάστευση πολύ περισσότερο α, στις δικές μας ε, τις χώρες, ε, στις αναπτυγμένες μας πόλεις. Πολύ περισσότερο από, ότι, από τις αναπτυσσόμενες αναπτυγμένες χώρες. Εμείς πηγαίνουμε στην Ινδία για να δουλέψουμε στις πόλεις της Ινδίας μαζί με τους, ε, με τους πρόσφυγες της Ινδίας για να οικοδομήσουμε τους θεσμούς κτλ. Υπάρχει μια αναπτυξιακή λοιπόν διάσταση στην ε, μετανάστευση. Το συμπέρασμα της έκθεσής μας ήταν ότι αν τη διαχειριστούμε καλά, είναι η φράση αυτή που χρησιμοποιούμε τώρα, θα ήταν πολύ σημαντική οικονομικά, πολιτικά, λόγω των δεσμών που θα δημιουργούσε μεταξύ των χωρών. Νομίζω ότι στο παρελθόν αυτό που κάναμε είναι να θεωρούμε ότι η μετανάστευση α, αναβοσβήνει με ένα διακόπτη. Τώρα τους φέρνουμε που έχουμε τις παχές αγελάδες και μετά τους διώχνουμε στις συχνές αγελάδες. Αυτό είναι ένα μεικτό μήνυμα που στέλνουμε και ο κόσμος καταλαβαίνει ότι πρόκειται για έλλειψη συνοχής εδώ στην πολιτική μας. Θα έπρεπε να κάνουμε μια ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ μετανάστευσης και προσφύγων. Ένα πιτσιρίκι 9 χρονών στο σχολείο είπε ότι είχε ένα φίλο ε, που ήταν παιδί πρόσφυγα. Και μου είπε ότι το γεγονός ότι κακομεταχειριζόμαστε του, τα παιδιά των μεταναστών, αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη ε, θεμητού εμπορίου και όχι ε, με, το ότι η μετανάστευση μας δημιουργεί προβλήματα. Όντω ε, υπάρχει μείωση των εμβασμάτων, αλλά τα εμβάσματα θα πρέπει να τα εντάξουμε στην αναπτυξιακή πολιτική για να τα επενδύουμε σωστά στις χώρες προέλευσης. Αλλιώ δεν υπάρχει σύνδεσμο κατά ανάγκη μεταξύ εμβασμάτων και ανάπτυξη. Αυτό το βρήκαμε από τι ε, έρευνε που κάναμε. Ε, το να συντονίσουμε τα πράγματα, ούτως ώστε οι αναπτυξιακές πολιτικές ε, χτίζουν σχολεία, κέντρα κατάρτισης ε, κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι πώς το διαχειριστούμε αυτό ως διαδικασία. Ένα άλλο θέμα που συζητάμε στην περιοχή μου είναι χρειαζόμαστε ξεκάθαρες πολιτικές ε, για την νόμιμη μετανάστευση, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τη λάθρο μετανάστευση και την παράνομη εμπορία. Επίσης, θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τα δικαιώματα των μεταναστών μέσω της νομοθεσίας και της εφαρμογής της νομοθεσίας. Να έχουν πρόσβαση στην υγεία, υγειονομική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση κτλ. Ε, Υπάρχει ένας νόμος τώρα που προστατεύει τους, ε, μετανάστες που χρησιμοποιούσαμε παλιά σε αγροτικές εργασίες, τους οποίους παίρναμε, τους στείδαμε και τους πετούσαμε. Θα πρέπει να τους φέρνουμε τους μετανάστες και να τους ενθαρρύνουμε συνεχεία να τους βοηθούμε να επιστρέψουν. για να υποστηρίξουν με την επιστροφή τους τις αναπτυξιακές μας πολιτικές. Να μην τους διώχνουμε απλώς. Το θέμα είναι να υπάρξει μια εταιρική σχέση για να υποφεληθούμε και η μεν και η δε. Για μια καλή σχέση μεταξύ βορρά και νότου. Έχουμε κάποια στοιχεία. Από το 2000 ε, για τους μετανάστες από το Μαλάουι. Προσπαθούμε μαζί με την ε, κυβέρνηση δηλαδή να συνεργαστεί με το Μαλάουι για να διπλασιάσει τον αριθμό των νοσοκόμων και να τριπλασιάσει τον αριθμό των γιατρών στις ε, δημόσιες υπηρεσίες του Μαλάουι. Να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα δυναμικό κατάρτισης Πού το πληρώνει ποιο, ο φορολογούμενο στην εκλογική μου περιφέρεια μεταξύ άλλων, να του δώσουμε επιμίστια στου μισθού στου γιατρού και στι νοσοκόμε, ούτω ώστε οι γιατροί αυτοί και οι νοσοκόμε να, να μείνουν εκεί. Επομένω έχουμε 40% περισσότερε νοσοκόμε και 50%, περισσότερες, περισσότερου γιατρού από ό,τι 4 χρόνια πριν. Επομένω δεν θα πρέπει τα πράγματα να τα βλέπουμε μονόπαντα. Ε, χρειαζόμαστε συνοχή και στις εθνικές μας πολιτικές. Γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα. Ε, δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των Υπουργείων. Κοιτάξτε, εμείς ε, εκπονήσαμε αυτό το θαυμάσιο ε, κείμενο, το οποίο δεν πέρασε, ας πούμε, σε κανένα άλλο Υπουργείο. Ε, αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο στην Βρετανία. Παντού. Και στις χώρες προέλευσης ακόμα. Ε, πώς όλες αυτές οι πολιτικές θα δημιουργούσε ένα συνεκτικό όλο. Επίσης, κάτι άλλο. Το πρόβλημα που έχουμε εμείς είναι ότι όχι δεν συνδέουμε την μετανάστευση με την ανάπτυξη, αλλά δεν συζητάμε καν για την ανάπτυξη. Εγώ προσπάθησα να πω στον Πρωθυπουργό μας ότι και η ώρα να μιλήσουμε για τη φτώχεια, για την ανεργία και να το θέσουμε στο κέντρο των, της ατζέντα μας της ε, οικονομικής. Να το αντιμετωπίσουμε ως πρόκληση αυτό. Όχι απλώς να στηρίξουμε τις τράπεζες. Αν το κάνουμε αυτό, θα μπορούσαμε να έχουμε μια διαδικασία που να οδηγεί στη συν-ανάπτυξη. Αυτέ είναι οι πραγματικέ σχέσει του 21ου αιώνα. Θα πρέπει να έχουμε διαφορετικέ οικονομικέ σχέσει, βιώσιμε. Να μην εξαρτώμαστε να μην παραμείνουμε στα στεγανά του 20ου αιώνα. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε τους φτωχούς στη μοίρα τους. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει, ποια θα είναι τα ωφέλη και για μας αν τα, τους βάλουμε τους ανθρώπους αυτούς στο κέντρο του οικονομικού μας σχεδιασμού. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ όσους πήραν το λόγο στο πάνελ. Ευχαριστούμε τους ομιλητές του πάνελ και τώρα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους που το ζήτησαν. Υπάρχουν δέκα ε, συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο, δέκα ομιλητές. Θα ήθελα να τους παρακαλέσω να μην περάσουν τα δύο λεπτά ο πρώτος είναι ο κύριος Μάξιμου, Μάξιμος Ζαραχόπουλος. Να επενέσω και εγώ την πρωτοβουλία της διοργάνωσης της ε, σημερινής συνδιάσκεψης. Το φαινόμενο της μετανάστευσης προς αναζήτηση καλύτερης ζωής θα εντείνεται όσο θα υπάρχουν άνθρωποι που πεινούν στην Ανατολή, τη στιγμή που στη Δύση δαπανούμε τεράστια ποσά στα Ινστιτούτα Δυνατίσματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας για τους οικονομικούς μετανάστες, η γυραιά Ήπειρος είναι παράδεισος σε σχέση με τις χώρες προέλευσής τους. Γι' αυτό, όσα μέτρα και αν ληφθούν, ακόμη και αν τα σύνορα της Ευρώπης φυλάσσονταν με ηλεκτροφόρα σύρματα, και πάλι θα είχαμε το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης. Τούτο δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να έχουμε καλύτερους και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς φύλαξης των ευρωπαϊκών συνόρων. Άλλωστε, η πατρίδα μου η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, είναι το σύνορο της Ευρώπης με την Ασία και η χώρα που δέχεται τη μεγαλύτερη ίσως μεταναστευτική πίεση. Το σημαντικότερο όμως, όπως είπε και ο κύριος Μαυρομάτης, είναι η αντιμετώπιση των αιτίων που οδηγούν στη μετανάστευση. Η εξάλληψη της φτώχειας και της πείνας, η ενθάρρυνση επενδύσεων και η δημιουργία προϋποθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης στις χώρες προέλευσης των οικονομικών μεταναστών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παγκόσμια οικονομική κρίση που δοκιμάζει τις αντοχές της οικονομίας των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελοχεύει νέες προκλήσεις και δημιουργεί νέα δεδομένα και για τη μεταναστευτική πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ένωση. Ο κίνδυνος επανεμφάνισης ενός κύματος ξενοφοβίας στην Ευρώπη το επόμενο διάστημα προβάλλει πολύ πιθανώς αν δεν αναλυφθούν έγκαιρα δράσεις. Ήδη χιλιάδες θέσεις εργασίας χάθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες και εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ζουν με τον εφιάλτη της ανεργίας. Ακραίες λαϊκίστικες φωνές δεν αποκλείεται να επιχειρήσουν ενεχοποίηση των μεταναστών για την αύξηση της ανεργίας. Άλλωστε, οι μετανάστες σε κάθε περίοδο ήταν ο εύκολος στόχος, όπως επεσήμανε το πρωί και ο κύριος Αμάνου. Πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε αυτόν τον κίνδυνο πιστεύω κλείνω κύριε πρόεδρε ότι θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στον αποτελεσματικότερο έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης και την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης στις τρίτες χώρες προκειμένου να συγκρατήσουν τους ενδυνάμει μετανάστες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Αρμάντο Φράνσα. Φράνκο. Η Φράντσα, λέει ο πρόεδρος, μάλλον δεν βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή. Η κυρία Μπονιβέρ από την Ιταλία. Βρίσκεται εδώ. Εδώ είναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η σημερινή συζήτηση διεξάγεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι αυτό στο οποίο αναφέρθηκαν και οι εμπειρογνώμονες, ε, όπως ο Jean-Pierre Garçon, ο οποίος κατήγγειλε μεταξύ άλλων ένα βαθμό υποκρισίας που υπάρχει όταν γίνεται λόγος για τη μετανάστευση. Θέλησε να μας υπενθυμίσει ότι η μετανάστευση στην Ευρώπη είναι ένα φαινόμενο που, σκοπό που μπορεί να αλλάξει την οικονομία μας, τις δημογραφικές μας τάσεις και τη δημοκρατία μας. Αυτό το φαινόμενο δεν μπορούμε εύκολα να το διαχειριστούμε. Και εμείς ως Ιταλοί είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε 4,5 εκατομμύρια μετανάστες από τρίτες χώρες. που συχνά έχουν φτάσει και στη δεύτερη ή τρίτη γενιά, έχουν κάνει παιδιά και εγγόνια. Ε, το βασικό πρόβλημα για την Ιταλία και για άλλες ε, ευρωπαϊκές χώρες είναι τι θα κάνουμε με την άφηξη των λαθρομεταναστών που αυξήθηκε το ποσοστό τους ε, κατά 60% το 2008 σε σχέση με το 2007 στην Ιταλία. Έχουμε ποικίλα προβλήματα λοιπόν τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Να μην ξεχνάμε ότι τα προβλήματα που συνδέονται με τη μετανάστευση μπορεί, μπορεί να οδηγήσουν σε κύματα ξενοφοβίας και το βασικό μας καθήκον είναι να τα ξεριζώσουμε εν το γεννάστε. Επίσης, γύρω από την χρηματοπιστωτική κρίση ε, πρέπει να πούμε τα πράγματα, ε, να τα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα ξεκάθαρα, να μην ομφαλοσκοπούμε. Οι μετανάστες είναι τα πιο ευάλωτα πλάσματα μέσα στις κοινωνίες μας και στις οικονομίες μας και θα είναι οι πρώτοι που θα χάσουν τη θέση τους, την εργασία τους. Πιστεύω ότι μια λογική πρόταση που γίνεται από την Διεθνή Τράπεζα, από την Παγκόσμια Τράπεζα, είναι να δημιουργήσουμε ένα ταμείο αλληλεγγύης για τους ευάλωτους, όπου θα πρέπει να στείλουμε το 0,7% των κονδυλίων που στέλνουμε για τις οικονομίες σε δυσκολία. Αυτό θα ήταν ένα θαυμάσιο πρόγραμμα και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να το σπρώξουμε, να το υποστηρίξουμε. Γιατί καλό είναι να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά μην ξεχνάμε και τους πιο φτωχούς πληθυσμού εντός αυτών. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα θα, δώσουμε, θα δώσω το λόγο στην κυρία ε, Καμπέλο Μαφούρο από το Λεσότο. Συγγνώμη, πρόκειται για έναν κύριο, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όταν άκουσα, α, όταν έλαβα την πρόσκληση αυτή, η πρώτη ερώτηση που έθεσε ήταν ποιος κάνει αυτή τη διοργάνωση και για ποιο λόγο. Γιατί τα θέματα τα οποία τίθεται εδώ ε, υπήρχαν πάντοτε. Γιατί γίνεται η διοργάνωση αυτή τη στιγμή. Νομίζω το πάνελ θα πρέπει να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Προσπαθώ να θέσω αυτό το θέμα γιατί πάντοτε μας κατηγορούν οι φορολογούμενοι ότι διοργανώνουμε υπερβολικά πολλά συμπόσια, συνδιασκέψεις κλπ. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα ότι δεν θα παραμείνουμε στα λόγια. Δεν θα είναι ακόμα ένα συμπόσιο ή μια συνδιάσκεψη και θα πεταχτούν τα έγγραφα στο σκουπίδο Ντενεκέ. Το ερώτημά μου είναι τι θα γίνει μετά, τι αναμένουμε ακριβώς από αυτή τη συνάντηση εργασίας. Κύριε Πρόεδρε, ξέρω ότι έχω μόνο δύο λεπτά στη διάθεσή μου. Αυτό το οποίο λέγεται συνήθως σε σχέση με τη μετανάστευση, ε, συνήθως αναφέρονται τα εμβάσματα. Ε, λέγον το επιχείρημα ότι τα χρήματα αυτά πηγαίνουν στη χώρα προέλευσης. Αν κάνει κανείς μια ανάλυση, ε, τα χρήματα αυτά, τα εμβάσματα πηγαίνουν μόνο στην οικογένεια, αλλά όχι στην ε, ανάπτυξη της χώρας η εκπαίδευση ενός ανθρώπου ε, χάνεται όμως. Ε, σκεφτείτε τι γίνεται με το AIDS, με τη φτώχεια κλπ. Ε, σκεφτείτε ποια είναι η κοινωνική κατάσταση στην Αφρική. Ε, χάνουμε τους εξειδικευμένους ανθρώπους. Ε, μιλάμε για το brain drain, τη διαφυγή εγκεφάλων ε, που πηγαίνουν ε, οι άνθρωποι αυτοί στην Ευρώπη και λοιπά, σε ανεπτυγμένες χώρες. Στην Αφρική θα τους ονομάζαμε ειδικού εμπειρογνώμονες. Αλλά πώς τους ονομάζουν στην ε, Ευρώπη, τους ονομάζουν μετανάστες. Έστω και αν τους χρειάζονται. Νομίζω ότι θα έπρεπε να επανεξετάσουμε αυτή τη σχέση γιατί αυτό το φαινόμενο διαρκεί εδώ και πολύ καιρό και τίποτα δεν γίνεται. Υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα, κύριε Πρόεδρε, όπως τα κοινωνικά δεδομένα για τις, των οικογενειών κλπ. κλπ. Καλά, κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω εδώ. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Καρλότο Μάργουες από την Πορτογαλία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Ανάπτυξης για τη διοργάνωση αυτής της συνδιάσκεψης, που νομίζω ότι έρχεται σε μια πολύ κατάλληλη στιγμή. Θα ήθελα να χαιρετήσω αυτή την πρωτοβουλία. Θα μας βοηθήσει στην ενεργειακή κρίση, την επιστημιστική κρίση, την οικονομική κρίση κλπ την κρίση αυτή συνήθως δεν αναφέρουμε, ενώ έχει μεγάλη σημασία σε στα μεταναστευτικά ρεύματα. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ των χωρών, αλλά και μεταξύ των διαφόρων υπήρων. Ορισμένες χώρες αποφάσισαν να λάβουν προστατευτικά μέτρα, αλλά νομίζω ότι εξαπατώνται γιατί χρειάζεται κανείς και βοήθεια απ' έξω για να επιβιώσει. Υπάρχουν 5 εκατομμύρια μετανάστες Πορτογάλοι που ζουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Πορτογαλία έρχονται και πολλοί μετανάστες. Για παράδειγμα, πολλοί κέρδισαν Ολυμπιακά μετάλλια χάρη της, για την Πορτογαλία και προέρχονται από την Αφρική. Και τώρα θα έρθω σε ένα σημαντικό σημείο. Οι επενδύσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι τρίτε χώρε είναι σημαντικέ. Ορισμένα προγράμματα που κάνουμε έχουν ξεκάθαρε κοινωνικέ και οικονομικέ επιπτώσει. Άλλα προγράμματα είναι θετικά ω προ την ανάπτυξη. Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να αναφερθώ σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ε, στην Γουινέα του Ισημερινού όπου για παράδειγμα γίνεται προσπάθεια να προστατευτούν τα τροπικά δάση και όπου οι πολίτες ε, εξοικειώνονται με την ε, σχετική προβληματική. Είναι εντυπωσιακό όταν μια χώρα που έχει τόσους, τόση ηλιακή ενέργεια όπως είναι η Αφρική να μην αξιοποιείται αυτή η ηλιακή ενέργεια. Ένας Ευρωπαίος βουλευτής αναφέρθηκε σχετικά. Ε, το, για παράδειγμα, ε, το μεσημέρι, στο μεσημεριανό διάλειμμα είδα την ετικέτα στο κρασί. Ε, δεν είδα εκεί να υπάρχει καμία βιολογική σήμανση, ενώ αντίθετα ε, μας είπαν ότι ήταν βιολογικά προϊόντα. Τώρα θα περάσουμε στον επόμενο ομιλητή, δημοσιογράφο, τον κύριο Πιμέντα, από την Πορτογαλία επίσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συγχαρώ και τον ΟΣΑ για αυτή τη συνδιάσκεψη, η οποία πράγματι διοργανώνεται σε μια συγκυρία όπου υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα ανάψη της ε, χρηματονομικής κρίσης. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι προκλήσεις είναι τεράστιες. Και ε, φαντάζομαι ότι στο εγγύς μέλλον θα, βρούμε, θα πρέπει να βρούμε κάποιους νέους τρόπους να βγούμε από την κρίση. Ξέρουμε ότι η μετανάστευση είναι συνιστά μια κοινή πρόκληση, έχει παγκόσμιες διαστάσεις και γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες και να παίρνουμε ε, πολιτικά μέτρα στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής με συνέπεια και συνεκτικότητα. Ο ΣΑ έκανε μια αξιολόγηση της μεταναστευτικής πολιτικής στην Πορτογαλία πριν από λίγο καιρό και είπε ότι η Πορτογαλία ε, έχει μια θετική μεταναστευτική πολιτική. Ε, η Πορτογαλία όπως υπόθηκε είναι χώρα που αποστέλνει πολλούς μετανάστες αλλά είναι και χώρα που υποδέχεται πλέον πολλούς μετανάστες. Γι' αυτό πρέπει να εφαρμόσουμε κάποιες σχετικές πολιτικές και χαιρόμαστε πάρα πολύ που όσα αξιολόγησε θετικά την δική μας μεταναστευτική πολιτική. Βεβαίως διατυπώθηκαν κάποιες συστάσεις προς την Πορτογαλία. Για παράδειγμα, ελέγχθη ότι η πορτογαλική κυβέρνηση θα πρέπει να συμπεριλάβει περισσότερο τους κοινωνικούς εταίρους στη χάραξη της μεταναστευτικής πολιτικής. Επίσης συνέστησε η Πορτογαλία να εντάξει καλύτερα τους μετανάστες, να τους εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης κλπ. Και επίσης θα πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα στους επιχειρηματίες. Βεβαίως διανύουμε μια κρίση, αλλά η Πορτογαλία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της ούτως ώστε να μπορέσει να εφαρμόσει τα αποτελέσματα του ΩΣΑ. Γιατί κύριε Πρόεδρε επιθυμούμε μια αλληλέγγυα και πολυπολιτισμική κοινωνία. Σε ευχαριστούμε πολύ.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 Έχουμε πολύ χαμηλό ΑΕΠ. Ε, κύριε Πρόεδρε, ε, χρειαζόμαστε πάρα πολλά δάνεια για να διατηρήσουμε την κοινωνική και οικονομική σταθερότητα και αυτό ε, δεν είναι εύκολο όταν κανείς επίσης πρέπει να εισαγάγει και την ενέργεια. Η χώρα μας είναι ιδιαίτερος ευάλωτη. Ποιες ελπίδες έχουμε με, μαζί με άλλες χώρες ε, για να μπορέσουμε να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Τι ελπίδες έχουμε όταν στο πλαίσιο των λεγόμενων εταιρικών συμφωνιών υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης. Μπορούμε να συμφωνήσουμε να αναλάβουμε κάποιες υποχρεώσεις να υπάρξει ένας ε, σεβασμός των θεσμικών αργάνων και να στραφούμε προς πράξεις και όχι λόγια. Τα βασικά θέματα, κύριε Πρόεδρε, είναι τα εξής. Ε, υπάρχουν παγκόσμιες ε, δεσμεύσεις για να υπάρξει ένας έλεγχος της μετανάστευσης. Υπάρχει η βούληση να υπάρχει η εσωτερική ισορροπία ποια συγκεκριμένα προγράμματα έχουμε μπροστά μας σαν οδικό χάρτη, τα οποία έχουν συμφωνηθεί παγκόσμια, ούτως ώστε να απορριφθούμε στην κρίση. Υπάρχει συνεκτικότητα και συνέπεια όσον αφορά τον έλεγχο της μετανάστευσης. Τι περισσότερο μπορεί να γίνει. Θέλουμε να κάνουμε αυτό το βήμα παραπέρα. Έχουμε το κουράγιο, κύριε Πρόεδρε, να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα και να ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος να, να βαγίσει το καράβι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Βίλιαμ. Χαίρομαι που οι ερωτήσεις σας επευθύνονται στο, στα μέλη του πάνελ. Προχωρώ με την κυρία Σαντάνα από την Ισπανία. Ευχαριστώ πολύ και σε ευχαριστώ που μας δώσετε την ευκαιρία να απευθυνθώ σε αυτό το φόρουμ. Εγώ προέρχομαι από τα Κανάρια και τα Κανάρια είναι μια περιοχή που γειτονεύει με τις αφρικανικές χώρες και εκεί έχουν ναυαγήσει πάρα πολλά πλοία μεταναστών και υπάρχουν τεράστιες διαφορές στο ΑΕΠ μεταξύ των χωρών. Είναι λογικό ε, τα Κανάρια να έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία προς το θέμα της μετανάστευσης. Ε, σήμερα έρχονται πολλοί μετανάστες σε εμάς και οι λόγοι είναι παρόμοια. έλλειψη ελευθερίας, φτώχεια κλπ. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να καταπολεμούμε αυτούς τους παράγοντες. Θα πρέπει να χαράξουμε ε, ολοκληρωμένες πολιτικές διαλόγου ε, σε, στις χώρες προέλευσης και στις χώρες υποδοχής. Γιατί υπάρχει μια συλλογική ευθύνη. Εγώ θα ήθελα να κάνω έκκληση προς το δίκαιο, ούτε ώστε στις χώρες όπου δεν υπάρχουν κανόνες δικαίου, όπου δεν υπάρχει το δίκαιο για να αντιμετωπίσουμε πιστούν τα προβλήματα της μετανάστευσης, ε, παράγονται φαινόμενα ε, κακομεταχείρισης των μεταναστών. Ε, η Ισπανική κυβέρνηση ηγείται αυτής της εκστρατείας. Θέλουμε να δεσμευτούμε ούτω ώστε να προσπαθήσουμε να απαλείψουμε το φαινόμενο της φτώχειας. Ελπίζω ότι η Ισπανική Προεδρία το πρώτο εξάμεινο του 2010 θα μπορέσουμε να επικυρώσουμε και πάλι τη στήριξη της Ευρώπης ως προς την επίτευξη των στοχών της χιλιετίας. Στην Ισπανία ε, δουλεύουμε σε δύο μεγάλα προγράμματα, ένα στρατηγικό πρόγραμμα ολοκλήρωσης και ένταξη όχι αυτών που φτάνουν στη χώρα αλλά αυτών που βρίσκονται ήδη εκεί και επίσης ένα νέο πρόγραμμα για την ε, πρόθεση της συνεργασίας το 2009 και 2010. Είμαι πεπισμένη ότι αυτή η οικονομική κρίση δίνει κάποιες ευκαιρίες για τη μείωση της φτώχειας και την επίτευξη του στόχου της ανάπτυξης δεν θα ήθελα να κλείσω παραλείποντας να πω ότι είμαι ικανοποιημένη που ζω στην ε, Ευρώπη όπου προστατεύουν τα δικαιώματά μου αλλά τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να κατοχυρώνονται για όλους τους πολίτες. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Σαντάνα. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Κέρες από την Πολωνική Γερουσία. Κέρες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, είμαι από την Πολωνία. Γίναμε μέλος το 2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με αρκετές άλλες χώρες. Θα συνεχίσω τώρα στα πολωνικά γιατί νομίζω ότι εκφράζομαι καλύτερα στα πολωνικά. Ε, το πάνελ ε, στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είπε ότι θα δει τα πράγματα της μετανάστευσης από την οπτική γωνία των κοινοβουλευτικών ε, εκπροσώπων. Εμείς είμαστε και εθνικοί βουλευτές και ευρωβουλευτές αλλά υπάρχουν και άλλα επίπεδα διακυβέρνηση σε περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας όχι μόνο στο κοινοβούλιο ή στη Γερουσία όχι μόνο στο κόρτε στην Ισπανία αλλά και στις περιφέρειές μας και στους νομούς μας και στις κοινότητές μας ένα ε, πρόβλημα που αναφέρθηκε είναι η μετανάστευση βορρά-νότου στη χώρα μου αυτή τη στιγμή α, αν αντιμετωπίζουμε και το πρόβλημα της ε, μετανάστευσης Ανατολής Δύσης και βλέπουμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μετανάστες ε, μετα... όχι μόνο από άλλες χώρες της, Ανατολ... της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από άλλες χώρες κυρίως από την Ανατολή Βιετνάμ, ε, Μεσαία Ανατολή κλπ. κλπ. Εκείνο που είναι σημαντικό λοιπόν είναι να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα αυτά και να πείσουμε και τις κοινωνίες μας να δεχθούν αυτά τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Ε, ερχόμενο σήμερα στη συνεδρίαση είδα μία αφίσα για μια διαδήλωση ε, για θέματα απασχόλησης, εργασίας, ανεργίας κτλ. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και πολλοί Πολωνοί πρόεδρε. Ωραία λέει ο πρόεδρος, η τελευταία ομιλήτρια είναι η κυρία Λίλ από τη Γερμανία. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ε, Λάλη είναι το μικρό μου όνομα, αλλά μπορείτε να με ονομάσετε έτσι. Ε, δεν, να με φωνάσετε έτσι, δεν έχω πρόβλημα. Θα ήθελα να σα επισημάνω το εξή. Η Γερμανία ε, έχει μία πεντηκονταετή ιστορία μετανάστευσης πίσω της. Και ε, θεωρούμε την μεταναστευτική πολιτική ως τμήμα της αναπτυξιακής πολιτικής. Αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Ε, θα ήθελα να σε επισημάνω δύο σημεία τα οποία αυτή τη στιγμή συζητιούνται στη Γερμανία. Από την πλευρά της κοινωνίας της υποδοχής υπάρχουν ε, οι εξή προσδοκίε του πληθυσμού. Λένε οι Γερμανοί πολίτε ότι οι γκάσταρμπάιτερ, οι ξένοι εργάτε, θα πρέπει να γίνουν κάποτε ισότιμοι πολίτε τη γερμανική κοινωνία όπως σας είπα, ξεκινήσαμε με τους λεγόμενους Gastarbeiter πριν από 50 χρόνια. Σήμερα μιλάμε για το φαινόμενο της κυκλικής μετανάστευσης και διαρωτώμε κατά πόσο δεν δίνουμε νέες ετικέτες σε παλιά δοκιμασμένα μοντέλα μετανάστευσης. Και νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα έπρεπε να σκεφτούμε κατά πόσο δεν, ε, δεν επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά τα σφάλματα της παλιάς μεταναστευτικής πολιτικής. Δεύτερον, όσον αφορά την ένταξη των μεταναστών. Οι άνθρωποι στις καινούργιες ε, χώρες ε, έχουν το μυαλό τους τραμμένο στην πατρίδα τους ε, θέλαν να τη βοηθήσουν και με τον τρόπο αυτό δεν έχουν καμία ενέργεια για να σωματωθούν οι ίδιοι στη νέα χώρα υποδοχή. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό οι καινούργιοι πολίτες σε μια χώρα να έχουν αυτό το αίσθημα ότι είναι πολίτες αυτής της χώρας και ότι εκεί βρίσκονται στο σπίτι τους και να μην έχουν πάντοτε κατά νου, πάντοτε ότι κάποια στιγμή θα επαναπατριστούν. Θα πρέπει νομίζω να εξεταστεί και αυτή η συνιστόσα του προβλήματος, κάτι το οποίο θεωρείται κάπως εγωιστικό από την πλευρά της χώρας υποδοχής. Αλλά ε, νομίζω ότι οι διακρίσεις κυρίως γίνονται όταν οι άνθρωποι δεν ενσωματώνονται καλώς στην ξένη κοινωνία. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα των διακρίσεων. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που μπέρδεψα το όνομα με το επώνυμό σας. Ο κύριος Ντέτον Τζόνσον που είναι μέλος του πάνελ θα πάρει το λόγο για να καταλήξει κάποια συμπεράσματα μέσα σε 12 λεπτά. Μάλιστα, δεν έχουμε και πολύ χρόνο ε, μπροστά μας για αυτό θα ήθελα να επιτρέψω αν θέλετε στους ομιλητές πήραν το λόγο πριν αλλά με αντίστροφη σειρά να δευτερολογήσουν αλλά δύο λεπτά μόνο ο καθένας ο κύριος Μπάτλ χωρίς μικρόφωνο α, προσπάθησα να περάσω το μήνυμα ότι αν θέλουμε να βρούμε στα στρατηγικές και λύσεις παγκόσμιες θα πρέπει να εντάξουμε τη μετανάστευση στις αναπτυξιακές μας στρατηγικές. Και το δεύτερο μήνυμα είναι αυτό που μόλις τώρα είπε η κυρία από τη Γερμανία. Είναι γεγονός ότι πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς υπηκότητα και ένα αίσθημα ότι είναι πολίτες. Η τραγωδία είναι ότι δεν έχουμε πρόβλημα με την ελεύθερη κυκλοφορία ε, εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή ε, χρήματος τέλος πάντων αλλά η ελεύθερη κυκλοφορία και μετακίνηση ανθρώπων δεν είναι το φόρτε μας πρέπει να σεβόμαστε την αξιοπρέπεια των ανθρώπων την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του μετανάστη και πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν δικαιώματα για όλους. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα για δουλειά και για να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους με ε, αξιοπρέπεια. Το θέμα βορρά-νότου είναι σημαντικό. Εμείς στο βορρά κοιτάζουμε αφιψηλού το νότο και αυτό είναι λάθος. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Διάρα, δύο λεπτά. Oui, merci. Euh, revenir un peu sur euh, beaucoup. Euh, Επανέλθω σε κάποια από τα ερωτήματα που ακούστηκαν από τους ομιλητές ε, στην αίθουσα σήμερα το πρωί και σήμερα το απόγευμα. Πολλοί είπαν ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτήν την υποκρισία σε ό,τι αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης της μετανάστευσης. Συμφωνώ απόλυτα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να, να θεωρούμε ως μείζον πρόβλημα και αίτιο για όλα μας τα προβλήματα τη, τη μετανάστευση. Θα πρέπει να δούμε τα θετικά της στοιχεία σε τοπικό επίπεδο όπως είπε ο κύριος Αποτολίτς, σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Θα πρέπει να δούμε τα θετικά στοιχεία της ε, μετανάστευσης για κάποιες χώρες. Εγώ με μεγάλη χαρά άκουσα α, κάποιους ομιλητές από χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ιταλία και η Ισπανία ακόμα που είπαν ότι ε, ήμασταν χώρες που στέλναν μετανάστες, ενώ τώρα είμαστε χώρες που υποδεχόμαστε μετανάστες. Το θέμα της μετανάστευσης είναι καθαρά οικονομικό και συνδέεται και με την ανάπτυξη. Στην Αφρική, ε, οι Αφρικανοί δεν φεύγουν επειδή τους αρέσει. Παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, την περίπτωση του Μαλή. Είναι βασικά οικονομικό το θέμα και συνδέεται με την αναπτυξιακή διάσταση και πολιτική. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε ε, ούτως ώστε η Ευρώπη και η Αφρική να έχουμε μία κοινή προσέγγιση στις ε, δημόσιες πολιτικές μετανάστευσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαυρομάτης, δύο λεπτά. Ε, θα απαντήσω απευθείας στον κύριο ε, Ματούρα από το Λεσότο, γιατί έθεσε δύο βασικά θέματα. Το θέμα κυρίως των εγκεφάλων, το θέμα των σχολείων δασκάλων και ένα κοινωνικό γενικότερα περιεχόμενο στην Επιτροπή Ανάπτυξης, τόσο στις δικές μου εκθέσεις όσο και οι άλλοι συνάδελφοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαστε σύμφωνοι ότι πρέπει να υπάρχουν σχολεία και δάσκαλοι στους τόπους από τους οποίους προέρχονται οι μετανάστες. Όταν υπάρχει σχολείο και δάσκαλοι πρέπει να ξέρουμε ότι μπορούν να μάθουν γράμματα και τα παιδιά, γιατί οι περισσότεροι είναι αναλφάβητοι και δυστυχώς δεν μπορούν να έχουν ούτε ενημέρωση διότι δεν υπάρχουν εφημερίδες και το μόνο μέσο που μπορούν να ενημερωθούν ή να ακούσουν είναι το ραδιόφωνο. Θα πρέπει να σας πω για τους εγκεφάλους. Εμείς παροτρύνουμε τις χώρες που υπάρχουν πραγματικά αξιόπιστα στελέχη, στελέχη πανεπιστημιακού επίπεδου να πηγαίνουν σε άλλες χώρες αλλά στη συνέχεια να επιστρέφουν από εκεί που προέρχονται, από τις χώρες δηλαδή που μεταναστεύουν. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι η Επιτροπή Ανάπτυξης ανέπτυξε μια μεγάλη δραστηριότητα στον τομέα των μίντια. Υπάρχουν σήμερα από τις ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως από προσπάθειες του BBC να έχουμε εκπαιδευμένους δημοσιογράφους οι οποίοι πηγαίνουν σε χώρες κυρίως της Αφρικής προκειμένου να στήσουν εφημερίδες, να στήσουν ραδιόφωνα και να εκπαιδεύσουν τους ντόπιου παράγοντες έτσι ώστε να έχουν ένα μέσο ενημέρωσης για να γνωρίζουν τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστώ. Ντάμπη προς τον κύριο από την Πολωνία. Ναι, τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να έχουν ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες για τη μετανάστευση. Δεν έχει νόημα να υπάρχουν ξενοφοβικές αντιμετωπίσεις. Ε, τα κοινοβούλια και οι βουλευτές πρέπει να είναι ανοιχτοί και να μπορούν να συζητήσουν ήρεμα, λογικά ε, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα θέματα της ε, μετανάστευσης και το ποια θα είναι η πολιτική που θα καταρτήσουν για το σχετικό θέμα. Τώρα, για τη μόνιμη για την κυρία από το Bundestag ε, για δίκαιο έχετε που ξεχωρίζετε τη μόνιμη μετανάστευση από τους Gastarbeiter ε, είναι όντως διαφορετικό πράγμα και βεβαίως η έννοια του Gastarbeiter μπορεί να είχε ή να έχει τη θέση στο διεθνές οικονομικό σύστημα αν θέλετε αλλά τώρα μιλάμε για τελείως διαφορετικό πράγμα ε, δεν μπορώ από την άλλη μεριά εγώ ε, να ζούσα στη Γερμανία τώρα θα ήμουν τρίτη γενιά ε, και θα με στέλνανε να πάω που στην Άγκυρα από την οποία ήρθε ο προπάπος μου νομίζω ότι ε, πρέπει να λάβουμε και ορισμένα τέτοια πράγματα υπόψη γι' αυτό μιλάμε για μόνιμη μετανάστευση κάποιοι μπορεί να θέλουν να γυρίσουν και οι άνθρωποι αυτοί βεβαίω, θα πάρουν την περιουσία τους και τα χρήματά τους θα γυρίσουν πίσω και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της χώρας από την οποία προήλθαν και ή μπορεί να γυρίσουν και να είναι πολύ καλοί γιατροί και να στήσουν εργαστήρια και νοσοκομεία στο Μαλί αλλά δεν μπορεί κανείς να πει στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά μεταναστών γύρνα πίσω απαραίτητο. Ε. Ναι, λέει ο κύριο Ντέιτον Τζόνσον. Θα ήθελα, επειδή έχουμε λίγο ακόμη χρόνο, να κάνω τρει τελικέ παρατηρήσει. Να υπογραμμίσω τρία πράγματα που μου φαίνονται σημαντικά. Στο αναφέρθηκαν τα κύρια ζητήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση και την ανάπτυξη εκτενώς αναφέρθηκαν τα εμβάσματα η διαρροή εγκεφάλων η διασπορά ο ρόλος της σε σχέση με τη, σε σχέση με τη βοήθεια κτλ τρία τρία όμως καινούρια πράγματα άκουσα εγώ σήμερα πρώτον ε, ε, θέματα συνέπειες και συνοχής και συνεκτικότητας των πολιτικών ε, ε, που μπορούν να συμπεριλάβουν θέματα μετανάστευσης και αναφέρθηκε εδώ ιδιαίτερα η ε, εμπορική πολιτική ε, και η ανάπτυξη των, η εμπορική πολιτική και η ανάπτυξη εμπορικής πολιτικής. Δεύτερο θέμα ε, αναφέρθηκε ότι, ότι υπάρχουν θεσμικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν έτσι, και σε διαφορετικά επίπεδα ε, διακυβέρνησης. Το επόμενο θέμα είναι κάποια ειδικά θέματα εγκατάσταση του μετανάστη, ε, απόκτηση υπηκότητας, πότε, πώς, υπό ποιους όρους κτλ. Και εδώ πράγματι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η αναπτυξιακή βοήθεια που δίνουμε έχει σαν στόχο να μειώσει την ανέχεια και τη φτώχεια. Από την άλλη μεριά η φτώχεια και η ανέχεια είναι το αίτιο για το οποίο φεύγει ο μετανάστης από τη χώρα του σε, πολλές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ε, αυτή η σχέση ίσως θα πρέπει να μελετηθεί λίγο παραπέρα και βεβαίως η, όπως ακούσαμε και αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα οι μετανάστες δεν είναι οι πιο φτωχοί των πιο φτωχών χωρών έτσι η διεθνής η μετανάστευση λοιπόν η, παγκόσμια μετανάστευση αν θέλετε και η παγκόσμια ανάπτυξη ε, συναρθρώνται με παράξενο τρόπο εδώ ε. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ο ρόλος των ανθρώπων της διασποράς. Ο κύριος Μαυρομάτης αναφέρθηκε σε νέες ιδέες βοήθειας ε, σε κάποιες, για κάποιες χώρες και αυτό που είπε ο κύριος Διάρα για το Μαλί είναι ένα καλό παράδειγμα. Η διασπορά είναι κάτι για το οποίο ε, είναι μια ομάδα ανθρώπων για τους οποίους ουσιαστικά δεν καταρτίζεται πολιτική πουθενά ούτε στη χώρα προέλευση, ούτε στη χώρα υποδοχής. Κάτι τι άλλο τώρα. Ο ρόλος των κοινοβουλίων τα κοινοβούλια θεωρητικά θα έπρεπε να είναι ο χώρος όπου κάποια προβλήματα βρίσκουν τη λύση τους. Φαντάζομαι ότι σε δια, για πολλά θέματα υπάρχουν κοινοβουλευτικές επιτροπές για το εμπόριο, για τη γεωργία, για την αλληλεία κτλ. Ε, αν, υπήρχε και, αν υπάρχουν αντίστοιχες επιτροπές μετανάστευσης, οι επιτροπές διασποράς, οι επιτροπές απόδημων αν θέλετε πολιτών ε, θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα και εδώ θα ήθελα να κλείσω το, το λόγο και να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ ε, Ευχαριστώ πολύ ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα τέσσερα μέλη του πάνελ Παρακαλώ να πάρετε τα καρτελάκια σας ε, με τα ονόματά σα. Λοιπόν, συντονιστής της επόμενης συνάντησης θα είναι ο κύριος Ξαβιέ Πράτς, που είναι διευθυντής Γενικής διεύθυνση Απασχόλησης. Ε, τα μέλη του πάνελ είναι ο κύριος Χουάν Φράιλε Καντών, η Σάρα Καν, η Μαρίζα Νταλρίμπλ Φιλιμπέρ και ο κύριος Κούντε Μαρτό.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 πιστεύουν ότι αυτό που αναμένεται από αυτούς είναι να, δώσουν μια, να συμβάλλουν στην ουσία του θέματος που συζητείτε. Αλλά ξέρετε και εγώ ξέρω ότι αυτό δεν είναι αληθές. Ο συντονιστής θα πρέπει να εξασφαλίζει οι ομιλητές να είναι ή δυνατόν σύντομοι για να έχει και το κοινό μια δυνατότητα να συμμετάσχει. Λοιπόν, Οκτώ λεπτά θα δώσω στον κάθε ομιλητή και θα είμαι πολύ αυστηρός όσον αφορά την τήρηση του χρόνου. Παρακαλώ να είστε σύντομοι στα σχόλιά σας. Αυτό θα είναι δύσκολο γιατί όπως ξέρετε το πάνελ αυτό πραγματικά προσφέρει μεγάλο ενδιαφέρον. Όταν εξάζουμε σήμερα τις αγορές εργασίας, αυτό το οποίο σκεφτόμαστε ε, ποια είναι η κατάσταση των αγορών εργασίας σήμερα. Είναι πραγματικά πολύ ε, πολύ άσχημη κατάσταση. Η Κομισιόν ε, θεωρεί ότι θα, μέχρι το 2010 θα χαθούν 6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Το 2010 ενδεχομένως τα ποστά αναργίας θα είναι 10%. Ενώ ορισμένε χώρε όπω η δική μου Ισπανία έχουν ήδη ξεπεράσει αυτό το ποσοστό ήδη σήμερα. Συνεπώ λοιπόν το θέμα τη αγορά εργασία είναι ένα θέμα που θέτει πολλέ προκλήσει. Και το θέμα είναι ποια θα είναι η μοίρα των μεταναστών σε αυτή τη συγκαιρία και πώς ε, μπορούν να συμβάλλουν στην ανάκαμψη και ενδεχομένως στην ε, ευημερία των χωρών μετανάστευσης. Θα δώσω το λόγο, χωρίς να καθυστερήσω, τώρα στον πρώτο ομιλητή, τον κύριο Χουάν Φράιλε Καντών, ο οποίος είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ενδιαφέρεται ιδιαίτερος για την τοπική διάσταση της μετανάστευσης. Κύριε Φράιλε Καντών, παρακαλώ να πάρετε το λόγο και να τηρήσετε τα 8 λεπτά χρόνο ομιλίας, αλλιώς θα διαμαρτυρηθώ. Ναι, θα προσπαθήσω να το κάνω. Θα παρουσιάσω το θέμα της ε, προσωρινής μετανάστευσης και πώς μπορεί να εισβάλλει στην ανάπτυξη και στη μείωση της παράνομης μετανάστευσης. Επίσης θα αναφερθώ στις ε, ενώσεις που δημιουργήθηκαν σε σχέση με τη μετανάστευση. Θα πρέπει καταρχήν να πούμε ότι το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι φαινόμενο ιδιαίτερος πολύπλοκο που προποθέτει διάλογο, διαβούλευση καθώς και ειδικέ δομές και μορφές συνεργασίας. Στην Ισπανία υπάρχει μια ολοκληρωμένη πολιτική μετανάστευσης μια πολιτική η οποία συμπεριλαμβάνει τις χώρες προέλευσης και διέλευσης και ε, ε, προορισμού. Προσπαθούμε να έχουμε μια ισορροπία με πρωτοβαλίες που μας ε, επιτρέπουν να διοργανώσουμε την, παράνομη, την νόμιμη μετανάστευση και να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση οι νόμοι μετανάστες θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με την αγορά εργασίας και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα απορρόφησης της αγοράς εργασίας. Συνεργαζόμαστε με τις ε, χώρες προέλευσης των μεταναστών ε, αναλύοντας τους στέτια της μετανάστευσης και προσπαθώντας να τα επηρεάσουμε. Επίσης προσπαθούμε να κάνουμε διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες ούτως ώστε τα προγράμματα προσωρινής μετανάστευσης να καλύπτουν τις ανάγκες της χώρας προορισμού, να μειώνουν τα φαινόμενα της παράνομης μετανάστευσης και να κατοχυρώνουν τα, ε, τα προνόμια των μεταναστών. Η προσωρινή μετανάστευση δεν είναι καινούριο φαινόμενο, ε, σημειώνεται εδώ και κάποιες δεκαετίες. Γι' αυτό το λόγο είναι βασικό να ορίσουμε ένα πολιτικό και νομικό ενδεδειγμένο πλαίσιο. Η Ισπανική νομοθεσία επιτρέπει να υπάρχει προσωρινή απασχόληση με διμερείς συμφωνίες ελέγχου των μεταναστευτικών ροών μεταξύ, ε, συμβάσεις που συνάπτουν μεταξύ Ισπανίας και χώρα προέλευσης. Αφορά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων από τη χώρα προέλευσης η επιλογή η οποία γίνεται στο επίπεδο των δύο διοικήσεων των χωρών με τη συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανισμών και τέλος η διαχείριση του συστήματος χορήγησης αδειών και θεωρήσεων στους εργαζόμενους παρόλο που είμαστε ικανοποιημένοι από αυτά τα αποτελέσματα, θέλουμε να βελτιώσουμε παρόλα αυτά τη λειτουργία αυτών των συμφωνιών και να αυξήσουμε την ποιότητα αυτών των διαδικασιών, να εγγυηθούμε την πλήρη εφαρμογή τη αρχή ε, ίση μεταχείριση, τη διαφάνεια και των μη διακρίσεων, να ενημερώνουμε του εργαζόμενου για τι δυνατότητε νόμιμη μετανάστευση, καθώ και για τι υποχρεώσει του και τα δικαιώματά του και επίση οι συμβάσει εξάλλου κάποιου μηχανισμού για να μειώσουν του κινδύνου τη παράνομη μετανάστευση, για να ε, τα, την παραποίηση των ε, εγγράφων και να μειώσουν την ε, παράνομη διακίνηση των ανθρώπων. Ε, με τον τρόπο αυτό αποφεύγουμε την οικονομική αποδιάρθρωση και οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνε για την πρόσληψη των εργαζόμενων. Με τον τρόπο αυτό ευνοούνται οι τοποθετήσει των ανθρώπων αυτών σε κατάλληλε θέσει. Και με τον τρόπο αυτό οι άνθρωποι αυτοί εισφέρουν με την εργασιακή του και κοινωνική του εμπειρία και επίση. Πολλέ φορέ με τον τρόπο αυτό οι επενδύσει αυτέ είναι παραγωγικέ. Από την άλλη, οι συμβάσει εγγυώνται την ε, ε, σωστή εφαρμογή των εργασιακών συμβάσεων. Ο εργοδότη είναι αυτό ο οποίο προτείνει πολλέ φορέ στέγη στου εργαζόμενου. Υπάρχει λοιπόν ένα διτό μηχανισμό, ο οποίο επιτρέπει επίση τον επαναπατρισμό και με τον τρόπο αυτό ε, διευκολύνεται ε, η παραμονή αλλά και η επιστροφή των εργαζόμενων στις χώρες τους. Το 2007 πάνω από 5.000 γυναίκες από το Μαρόκο ήρθαν στην Ισπανία χωρίς ειδίκευση ε, και εργάστηκαν σε αγροτικές ε, καλλιέργειες. Λοιπόν, οι μηχανισμοί αυτοί δίνουν στους εργοδότες το κατάλληλο εργατικό δυναμικό που έχουν επαγγελματική εμπειρία και διευκολύνουν την ένταξή τους στην εργασία. Ε, κλείνοντας θα ήθελα να, σας, να αναφερθώ σε μια πρακτική η οποία απαντάται στο εγχειρίδιο ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το εγχειρίδιο για την ε, θέσπιση ε, εργασιακών ε, πολιτικών απασχόλησης συγγνώμη, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ανάπτυξης στην Καταλανία που απευθύνεται σε εργαζόμενους προσωρινής απασχόλησης. Αφορά και επιλέγονται εργαζόμενοι οι οποίοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη της κοινότητας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε και για το ότι σεβαστήκατε το χρόνο. Η κυρία Σέρα Κάν, που είναι από το Όσλο, επί έξι χρόνια ήταν μέλος του Συμβουλίου των τοπικών αρχών του Όσλο ασχολήθηκε είναι και μέλο του Κοινοβουλίου, ασχολήθηκε με θέματα μεταναστών, μπορεί να μας πει πολλά πράγματα για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και να μας πει και το πώς αντιμετωπίζονται οι άντρες σε σχέση με, τους, με τις γυναίκες. Ε, σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας, πολύ κολακευτική. Ε, σας ευχαριστώ που μου δώσατε το, την ευκαιρία να έρθω εδώ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εκδήλωση στις Βρυξέλλες ιδιαίτερα για μένα, γιατί τώρα στο Όσλο κάνει πάρα πολύ κρύο, χιονίζει ασταμάτητα. Επομένως, μου φαίνεται πραγματικά ότι έχει κοινικά καύματα εδώ στις Βρυξέλλες. Οι κοινωνίες μας αλλάζουν ε, και η αγορά εργασία λόγω της μετανάστευσης. Ε, Ιδίω ε, σε ό,τι αφορά τα δύο φύλλα, η μετανάστευση ε, είναι ένα καυτό θέμα και στις ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ τα βλέπω τα πράγματα ως την Νορβηγίδα, αλλά ξέρω πολύ καλά τι γίνεται γενικά σε όλες τις σκανδιναβικές χώρες. Σουηδία, Δανία κτλ. Ε, έχουμε όλοι παρόμοια εμπειρία με τη μετανάστευση. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται με τη μετανάστευση των γυναικών και των παιδιών επίσης. Ε, άλλη είναι η εμπειρία στις ΗΠΑ, άλλη είναι η εμπειρία στο ΗΠΑ. Έχουμε μετανάστες δύο γενεών. Τώρα φτάνει και το τρίτο κύμα, η τρίτη γενιά. Οι πρώτοι μετανάστες φτάσαν στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70. Τέλειωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Εμείς χρειαζόμαστε φθηνό εργατικό δυναμικό ε, στα εργοστάσια μας για να χτίσουμε τις υποδομές μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν φθηνά εργατικά χέρια και όσοι ήρθαν ήταν ε, εργάτες από το Πακιστάν, την Τουρκία, την Ινδία, που ήρθαν στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο στα δεκαετία του 50 και του 60, αυτά στην Ευρώπη. Τότε ήρθαν μόνο άντρε. Δεν πιστεύαμε ότι θα έρθουν και θα παραμείνουν στην Νορβηγία. Εμείς τους δώσαμε φθηνέ δουλειές στην Νορβηγία και δεν, είχα, δεν τους ζητήσαμε τίποτα. Δεν τους είπαμε να μάθουν τη γλώσσα μας, να εκπαιδευτούν, να αποκτήσουν ειδίκευση και προσόντα, γιατί στην ε, τότε νοοτροπία μας αυτοί οι άνθρωποι ερχόταν να δουλέψουν, να κερδίσουν λεφτά και να επιστρέψουν μετά από, μετά, μετά από 5, 6, 7 χρόνια. Αλλά όμως δεν έφυγαν. Πήγαν στο Πακιστάν και στην Τουρκία, παντρεύτηκαν και συνεχεία έφεραν και τις γυναίκες τους στην ε, Νορβηγία. Και πολύ καλά έκαναν, γιατί έτσι γεννήθηκα και εγώ. Το πρόβλημα ήταν ότι πολλές από αυτές τις ε, γυναίκες όμως είναι αγράμματες, δυστυχώς. Επομένως, αυτή είναι η νέα γενιά φτωχών στην Ευρώπη. Από εκεί προέρχονται, από αυτό το περιβάλλον. Τώρα έχουν παιδιά. Έχουμε φτάσει στη δεύτερη γενιά λοιπόν μεταναστών, στην Νορβηγία τουλάχιστον. Και δυστυχώς πολλά από τα κορίτσια δεν μπορούν να πάνε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πολλά από τα κορίτσια αναγκάζονται να παντρευτούν νωρίτερα. Πολλά αγόρια φεύγουν από το σχολείο ε, ασχολούνται με κλιματικές δραστηριότητε, φυλακίζονται εν συνεχεία. Επομένως, είχαμε μεταναστευτικές πολιτικές, οι οποίες δεν θα έλεγα είναι εντελώς ανεπιτυχείς, αλλά ε, τους έλειπαν πάρα πολλά στοιχεία. Επομένως, δεν σκοπεύαμε να... Ούτε είχαμε καμιά πολιτική για να εκπαιδεύσουμε αυτά τα παιδιά που μεγάλωναν στην Νορβηγία. Δεν είχαμε εργατική πολιτική για αυτά τα παιδιά. Τώρα κάνουμε μια προσπάθεια. Το πρόβλημα είναι ότι όταν περιμένεις πάρα πολύ με τους μετανάστες, σου κοστίζει. Σου κοστίζει πολύ περισσότερο από ότι αν έχεις μια προληπτική πολιτική. Τώρα στην Νορβηγία χρειαζόμαστε περισσότερα εργατικά χέρια λόγω της χρηματοπιστωτική κρίσης. Τώρα προσπαθούμε να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη με αυτά του παρελθόντος. Έχουμε προγράμματα κατάρτισης για όσους φέρνουν τις γυναίκες τους ή, τα παιδιά, ή τους άντρες τους ε, στην Νορβηγία για να δουλέψουν αγορά εργασία στην Νορβηγία. Προσπαθούμε να έχουμε μια καλή μεταναστευτική πολιτική για τα παιδιά. Γιατί μόνο τότε θα υπάρξει κοινωνική συνοχή. Ένα άλλο θέμα για την κοινωνική συνοχή είναι πώς θα τα καταφέρουμε να συνεπάρξουμε όταν έχουμε διαφορετικές κουλτούρες και θρησκείες. Πώς θα καταφέρουμε να συνεπάρξουμε. Στη Γαλλία έχουμε ένα μη θεοκρατικό κράτος. Κανένας δεν μπορεί να, φορά, να φέρει δημοσία ε, θρησκευτικά σύμβολα. Αλλά ακόμα ε, στην Νορβηγία υπάρχει το καθεστώς της Εκκλησίας. Σήμερα στο Όσλο, στην Νορβηγία γενικά, γίνεται μια τεράστια συζήτηση για το αν θα επιτρέψουμε στους αστυνομικούς ε, άντρες και γυναίκες στην Νορβηγία να φοράνε το φουλάρι. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση. Ε, λένε ότι στη Βρετανία γίνεται αυτό. Η αστυνομία του Λονδίνου το επιτρέπει. Αλλά εμεί το αντεπιχείρημα είναι ότι ο αστυνομικό θα πρέπει να είναι μια ουδέτερη φιγούρα γιατί α, πρέπει να επιλύσει συγκρούσεις. Και με το χιτζάπ, με αυτό φουλάρι, δίνουμε το λάθος μήνυμα. Έχουμε πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, πολλές και δύσκολες. Αναφέρατε τώρα το φύλλο και τη μετανάστευση. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Ποιοι χάνουν σε αυτές τις συζητήσεις για τη μετανάστευση. Είναι οι φτωχοί, οι γυναίκες και τα παιδιά. Τα, και τα καταφύγια ε, γυναικών ε, στην Νορβηγία υποδέχονται πάνω από το 80% κυρίως μετανάστριες και πάνω από το 80% είναι ε, άνεργες ε, στο Όσλο αυτές οι μετανάστριες. Αυτές που δεν εμφανίζονται στα προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας είναι γυναίκες. Είναι πραγματικά επώδυνο να μιλάμε για αυτά τα θέματα, γιατί δεν θέλουμε να είμαστε ρατσιστές. Και δεν θέλουμε να μιλάμε για αυτά τα ακαθόδη θέματα τη μετανάστευση. Κι όμω πρέπει να μιλήσουμε δυνατά και για τη μετανάστευση και για τι γυναίκε. Γιατί έχουμε μια ευθύνη απέναντι σε αυτές τις γυναίκες που φτάνουν στι δυτικές χώρε. Γιατί μιλάμε με τέτοια ευκολία για τη Σαρία και για τις γυναίκες στο Ιράν, αλλά όταν αυτές οι γυναίκες έρχονται στην ε, Νορβηγία, ε, στη Σουηδία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, φοβόμαστε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, για τον Ισλαμικό νόμο. Μία ερώτηση προς τους υπόλοιπους ε, ομιλητές του πάνελ, την οποία θα υποβάλω όμως αργότερα. Νομίζω ότι είπα αρκετά και θα, και θα κρατήσω λίγο χρόνο για να παρέμβω εκ νέου μετά. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τόσα είπατε. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στην επόμενη ομιλήτρια που είναι από τη Τζαμάικα. Ε, εσείς παραπονηθήκατε για τον καιρό. Αυτή νομίζω ότι εκεί θα έχει να μας πει καλά πράγματα για τον καιρό. Η κυρία Μαρίζα Νταλίμπλ Φιλιμπέρ που είναι νομικός, εκπρόσωπος του Εργατικού Κόμματος, βουλευτής θα ξέρετε πολύ καλά, θα μιλήσετε φαντάζομαι για το θέμα των φύλων και επίσης για τις χώρες και τους πληθυσμούς που έρχονται στην Ευρώπη. Κυρία μου, λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί φίλοι, είναι πάρα πολύ ωραίο που βρίσκομαι εδώ στις Βρυξέλλες. Εγώ δεν έρχομαι από κρύα χώρα ε, αντιθέτως εδώ μου φαίνεται ότι κάνει κρύο εμένα στην ε, Τζαμάικα ε, είναι τροπικός ο καιρός αλλά φε, έχουμε ήλιο και αυτό δεν αντικαθίσταται εύκολα λοιπόν να σας πω μερικά πράγματα για τη μετανάστευση από την οπτική γωνία της Τζαμαϊκά. Η μετανάστευση είναι αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας αν θέλετε της Τζαμάικα. Ξεκινήσαμε από το σκλαβεμπόριο, μετά ε, ε, εισαγωγή αν θέλετε άλλων εργαζομένων ή ατόμων όταν δεν υπήρχε πια σλαβεμπόριο και μετά ε, άρχισαν η, η Τζαμαϊκά να στέλνει κόσμο που είχε ε, κάνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ε, τη δεκαετία του 40 ε, προ, στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, για να αντιμετωπιστούν τα οι ανάγκες μετά τον πόλεμο επόμενη φάση αν θέλετε της μετανάστευσης ήταν στη δεκαετία του 60 όπου οι συμπατριώτες μου έφευγαν από, ε, δεν πήγαιναν πια στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά στις Ηνωμένε Πολιτείες ή εν πάση περιπτώσει στην ε, Βόρεια Αμερική όμως η συμπατριώτες μου συνεχίζουν ακόμη και τώρα που έχει σταματήσει μεγάλη φυγή αν θέλετε να συνεχίζουν να πηγαίνουν στην, στις Ηνωμένε Πολιτείες, στο Καναδά, στη Βόρεια δηλαδή Αμερική ενώ οι μετανάστες που πάνε στην ε, Ευρώπη είναι ελάχιστοι είναι της τάξης του 2% των συνολικών μεταναστών που φεύγουν από τη χώρα μας μιλάμε επίσης για την ε, ε μιλάμε επίσης ε, για μετανάστες τώρα που φεύγουν από την Τζαμάικα αλλά με πάρα πολλά προσόντα και ικανότητες στη δεκαετία του 90 ήταν ε, ελεύθεροι επαγγελματίες ε, management και δεν ξέρω τι ε, γιατί διότι οι πολιτικές μετανάστευσης των χωρών όπου πήγαιναν οι Τζαμαϊκανοί δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά απαιτούσαν κάτι τέτοιο η στον τομέα της υγείας και της παιδείας ε, ε, οι Τζαμαϊκανοί ε, και είναι πραγματικά ε, ε, εργάζονται σημαντικά και καλά στους τομείς αυτού στο εξωτερικό έφευγαν λοιπόν από την Τζαμάικα συμπατριώτες μας με προσόντα και πήγαιναν σε άλλες χώρες και έτσι άρχισε να δημιουργείται στην Τζαμάικα ένα κενό σε νοσηλεύτριες, γιατρούς, δασκάλους κτλ στον τομέα των υπηρεσιών επίσης άρχισε να δημιουργείται ε, μια αντίστοιχη κίνηση ε, οι Τζαμαϊκανοί πηγαίνουν στον, για τον τριτογενή τομέα ε, στην, στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι τόσο πολύ στον Καναδά Α, και δημιουργούνται με αυτή την έννοια τα κενά στη χώρα μας. Συγχρόνως βεβαίως η μετανάστευση, η τάση μεταναστευτική των, ε, των Τζαμαϊκανών που φεύγουν μειώνεται, αλλά παρόλα αυτά ε, υπάρχει πρόβλημα. Η ανα... Τώρα για τα φύλλα η στη δεκαετία του 70 είχαμε μία διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών της τάξης του 7% του 3,5% με συγχωρείτε ε, τώρα ε, είμαστε στο 7% ε, βλέπουμε και άλλου είδους διαφορές ε, αντίστοιχες, ανισότητες αντίστοιχες ε, και στον ε, τομέα της παιδείας και βεβαίως αυτό επηρεάζει αργότερα και τους ρόλους των φίλων και τις ε, και βεβαίως όλα αυτά αυτά οφείλονται εν πολλής στην κουλτούρα της χώρας μου η οποία αποδίδει ε, διαφορετικούς ρόλους στον άνδρα και στη γυναίκα οι οποίοι από εκεί και πέρα γίνονται ε, αποδεκτή και στο εξωτερικό. Ε, τα πράγματα βεβαίως έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια σε σχέση με πολύ παλιότερα και η γυναίκες, τα κορίτσια ε, εκπαιδεύονται καλύτερα και φεύγουν συγχρόνως από τη χώρα μας, από την πατρίδα μου πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Η χώρα μου λοιπόν αυτή τη στιγμή ε, η πλήττεται αν θέλετε από το φαινόμενο αυτό της διαρροής εγκεφάλου και βεβαίως ε, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ε, σημαντικά ο αριθμός των εμβασμάτων που παίρνουμε από το εξωτερικό γύρω στα 2 δις δολάρια το χρόνο όμως λόγω της οικονομικής κρίσης την οποία διατρέχουμε ε, αυτή τη στιγμή όλοι μας ήδη έχουν αρχίσει τα εμβάσματα να πέφτουν ε, επίσης υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στην φροντίδα των παιδιών, των μικρών παιδιών και έχουμε φτάσει στην κατάσταση ο κύριος ε, γονιός το, το κύριο άτομο το οποίο φέρνει χρήματα στο σπίτι να είναι οι γυναίκες πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα εμβάσματα αυτά ε, και πώς χρησιμοποιούνται και πού χρησιμοποιούνται όταν φτάσουν στην Τζαμάικα αν χρησιμοποιούνται μόνο για την επιβίωση, την ε, κατανάλωση, την απαραίτητη, την καθημερινή της οικογένειας ή αν χρησιμοποιούνται για, την να σας πω, επένδυση, για επενδυτικούς σκοπούς. Σε Τα τελευταία χρόνια εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης ε, και πραγματικά το πρόγραμμα αυτό είχε αρκετές επιτυχίες και κάποια σχέδια αρκετά ενδιαφέροντα για την περιφερειακή μετανάστευση υπάρχουν τώρα και άλλα προγράμματα που εφαρμόζουν που εφαρμόζονται ε, σε συνεργασία με τις Ηνωμένε Πολιτείε και τον Καναδά και πολλοί από τους συμπατριώτες μου ε, σε, άλλες, σε άλλα νησιά της Καραϊβικής ε, ασχολούνται με τα ε, σχέδια αυτά, με τα προγράμματα αυτά και πραγματικά είδαμε ε, βλέπουμε ότι γενικότερα στην Καραϊβική αλλά και στη δική μου τη χώρα ε, για σε πολλές περιπτώσεις τα κενά που δημιουργήθηκαν από τη διαρροή εγκεφάλων για ειδικά καταρτισμένα άτομα με ψηλά προσόντα καλύπτονται από άλλους, ε, από ξένους αλλά πάντα από την Καραϊβική παραδείγματος χάρη από την Κούβα. Και πολλοί ζητούν ε, δουλειά στη χώρα μου και το βλέπουμε από αυτούς που απαντούν στις μικρές αγγελίες όταν προκυρήσουν θέσεις εργασίας. Κλείνοντας να πω ότι το θέμα της μετανάστευσης είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και χρειάζεται πολλές περαιτέρω μελέντες για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί και ποιες είναι οι πιθανές λύσεις. Χαιρόμαστε που η Τζαμέικα ε, επελέγει ως μία χώρα στόχος για το πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο έχει σε στόχο να εξετάσει ε, σε μεγαλύτερο βάθο βάθος το φαινόμενο της μετανάστευσης. Πραγματικά με ανυπομονησία περιμένουμε να ακούσουμε ε, και άλλες συζητήσεις και ερωτήσεις αν υπάρχουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ ε, που μας ε, αναφερθήκατε στις γυναίκες της Τζαμάικα και μας είπατε ότι παίρνουν την εκπαίδευση και την εργασία πολύ σοβαρότερα από τους άνδρες και έχουμε πολλούς δείκτες που μας δείχνουν ότι οι γυναίκες στην Τζαμάικα ε, εξισώνονται με τις γυναίκες στην Ευρώπη. Τώρα, ο τελευταίος ομιλητής μας είναι ο κύριος Κόντε Μαρτό, ο οποίος εργάζεται σε μια εταιρεία DHL, μια γνωστή σε όλους μας ε, εταιρεία και ο οποίος ε, έχει γράψει άρθρα σχετικά με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και θα παρουσιάσει τη μετανάστευση ε, από το οπτικό πρίσμα της ε, πολυεθνικής συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Είμαι δεύτερος ομιλητής από το χώρο των επιχειρήσεων και κάθομαι στην ίδια θέση. Είναι η θέση business στην αίθουσα αυτή. Λοιπόν, ε, ποιο είναι ο ρόλος μου στην DHL. Είμαι επικεφαλής της, ε, της υπηρεσιών στην Ευρώπη. Αγοράζω μάλλον υπηρεσίες και κυρίως ε, υπηρεσίες ε, και ε, ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για τις τάσεις της ε, εξέλιξης γιατί φαίνεται ότι αντιμετωπίζουμε και εμείς τα ίδια προβλήματα αλλά τα εξετάζουμε κάτω από μια διαφορετική οπτική γωνία. Εμείς ως Deutsche Post είμαστε παρόντες σε πάνω από 200 χώρες ε, στην Ευρώπη και απασχολούμε 500.000 άτομα και υπάρχουν ένα ή δύο άτομα τα οποία απασχολούνται άμεσα μέσω τρίτων μερών. Και αυτό σημαίνει ότι τριπλασιάζεται το προσωπικό μας. Συνεπώς έχουμε ε, μια ε, τεράστια επιρροή στα όσα συμβαίνουν. Ε, τώρα, ενημερωτικά, θα ήθελα να σας πω να σα κάνω μια παρουσίαση που δίνει μια συνολική εποπτεία. Δεν είμαι απολύτως ειδικό να το κάνω. Ε, συνήθως ε, είναι κάποιοι από τους βοηθού μου που το κάνουν σε δύο ή τρία λεπτά αυτή την παρουσίαση. Εγώ χρειάζομαι πολύ περισσότερο χρόνο, τρεις ε, ώρες. Εμείς ασχολούμαστε με όλα τα επίπεδα, με διαφόρους τύπους δεξιοτήτων. Ε, Είμαστε πολυεθνικοί όπως σας είπα και ε, έχουμε δημιουργήσει μια ταυτότητα της εταιρείας μας η οποία πραγματικά διευκολύνει τα πράγματα για τους μετανάστες οι οποίοι αποκόβονται από την εθνική του ταυτότητα και συνδέονται με ένα καινούριο κόσμο, ένα κόσμο ο οποίος έχει μια πολύ ξεκάθαρη επωνυμία, Deutsche Post. Είναι ιδιαίτερος αναγνωρίσιμο λοιπόν. Και θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα, κάτι το οποίο άκουσα νωρίτερα σήμερα. Η, η, με ε, σε μια χώρα, Κάποιος μου είπε στη Μασαλία ότι μια κυρία πήγε από την ε, Μπρετάνια στην ε, Μασαλία. Ε, δηλαδή έκανε μια απόσταση χιλίων χιλιόμετρων. Και παραμένει μια γαλίδα επίκοος. Είναι παράδοξο ότι ε, στην, μέσα στην Ευρώπη ακόμα υπάρχουν τα σύνορα μεταξύ των χωρών. Εμείς ε, έχουμε πάρα πολλές διαφορετικές υπηκότητες, ανθρώπους από ολόκληρο τον κόσμο και το συνεκτικό στοιχείο είναι ακριβώς αυτή η ταυτότητα της εταιρεία. Παρόλα αυτά υπάρχει μια νέα ε, γενιά και όταν εγώ έκανα ε, την πρόσληψη του, της Ευρωπαϊκής Ομάδας, διαπίστωσα ότι σε μια ομάδα οκτώ ατόμων, πέντε από αυτούς ανήκουν σε μια γενιά που λένε ότι παντού όπου γη και πατρίς. Και πραγματικά έχουν ένα πολύ καλό επίπεδο εκπαίδευσης είναι άνθρωποι που έχουν πολύ καλή κατάρτιση. Εμείς φροντίζουμε να τους εκπαιδεύσουμε ακόμα περισσότερο. Είναι ιδιαίτερα ευέλικτοι όσον αφορά τους ρόλους που αναλαμβάνουν. Και συνήθως είναι γυναίκες οι άνθρωποι αυτοί. Ε, κοιτάζοντας τη σύνθεση της ομάδας μου, κοιτώντας την ομάδα μου μάλλον, η ζωή μου γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Τώρα, ένα από, τα, από τις ερωτήσεις που εμφανίζονται συχνά στις συνεντεύξεις είναι ε, μια γυναίκα που έρχεται από το Βιετνάμ. Όταν τη ρώτησε για τα κίνητρά της, ε, της είπα πόσο δύσκολο είναι για μια νέα γυναίκα από το Βιετνάμ να εργάζεται σε μια γερμανική εταιρεία προσπαθώντας να αποδείξει ότι είναι εξίσου ικανή να ανέλθει μέχρι το επίπεδο του management. Αυτό ισοδυναμεί με ένα αίτημα μια ανάπτυξης. Ε, το κοινό κίνητρο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ε, δεν έχουν ρίζες. Ε, σπίτι τους είναι όλος ο κόσμος και θέλουν να αναπτυχθούν περισσότερο, να αναπτυχθούν ήδη σαν προσωπικότητες και να αναλάβουν ευθύνες. Εάν δείτε αριθμού και στατιστικά νούμερα, όλα αυτά είναι ωραία. Αλλά μοιάζουν σαν αερολογίες. Όταν κανείς μιλάει πρόσωπο με πρόσωπο με ένα άτομο, μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι γίνεται. Και πρόκειται πράγματι για μια γενιά η οποία θα οικοδομήσει το μέλλον. Γιατί για την εταιρεία μας είναι μια ευκαιρία. Όταν, αυτοί είναι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούμε όταν δημιουργούμε νέα κέντρα, νέα αισθητούτα κατάρτισης. Και είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τα ημεία στην εταιρεία μας. Και και γιατί έχουν ακριβώς αυτό το κίνητρο της ε, ανάπτυξης ολοκλήρωσης της προσωπικότητάς τους και της ανέλυξης. Βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι γιατί μια εταιρεία πρέπει να είναι αρκετά στέρεη για να μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, για να είναι σε θέση να κάνει αυτό που κάνει μια εταιρεία. Ε, και πρέπει ε, να υπάρχει η έννοια του το ανήκει κανείς σε μια ε, παγκόσμια εταιρεία, σε μια πολυεθνική εταιρεία. Εδώ οι ξεκάθαρες αξίες βοηθούν, ο δοντολογικός κώδικας επίσης εφόσον είναι ξεκάθαρος μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος γιατί η εταιρεία μας αντανακλά είναι καθρέφτης της κοινωνίας, καθώς και τα προβλήματά της. Γιατί από την άλλη έχουμε μια πολύ ανοιχτή ατμόσφαιρα, πολυπολιτισμική, ε, έχουμε ένα πνεύμα συναδελφικότητας. Συνεπώς, για μας υπάρχει μια μεγάλη ευελιξία και με τον τρόπο αυτό αναπτυσσόμεθα σαν μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες. Εμείς δεν παράγουμε τίποτα, παρέχουμε υπηρεσίες και αυτό βέβαια μας καθιστά κάπως τροτούς. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μία εμπειρία, μία ε, υποχρέωση και χρειαζόμαστε πραγματικά ικανότητες, ταλέντα. Και νομίζω ότι πολλοί από τους ε, μετανάστες έχουν αυτές τις ικανότητες. Επίσης χρειαζόμαστε σε επενδύσεις. Αυτό είναι κάτι που οι πολυεθνικές εταιρείε μπορούν να το κάνουν καλύτερα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορούμε ακόμα και σε σκληρές εποχές, μπορούμε να βάλουμε στην άκρη κάποια χρήματα να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη. Επίσης συνεργαζόμαστε με κυβερνήσεις. Το κάναμε ήδη με την γερμανική κυβέρνηση αλλά και με κυβερνήσεις άλλων χωρών και με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, όπως είπε και ο συνάδελφος από τη Manpower, είναι ότι κρίνουμε ανάλογα με τις συνθήκες, με τη συγκυρία. Βεβαίω υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι και ο βασικότερος κίνδυνος είναι η μη εναρμόνιση των πολιτικών σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένας άλλος κίνδυνος είναι το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις καθορίζονται από την Wall Street και κανείς ζούμε όλοι σε έναν πλασματικό, σε έναν εικονικό κόσμο αλλά όπου τα προβλήματα είναι πραγματικά και όλες οι χώρες επενδύουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα αλλά κανείς δεν γνωρίζει που θα πάνε αυτά τα χρήματα. Συνεπώς λοιπόν υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Μπορούν οι χώρες και οι κυβερνήσεις μπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη νέα γενιά. Ορισμένοι είπαν ότι αυτό είναι φυκτό. Αλλά αυτό θα γίνει ίσως μέσω της ανάπτυξης. όσον αφορά το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων, πράγματι υπάρχει, υφίσταται αυτό το φαινόμενο, αλλά υπάρχει, εμείς προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη των εγκεφάλων. Ε, και συνεχώς υποστηρίζει ο κάθε μάνατζερ ένα ή δύο τρία στελέχη της ομάδος του, ώστε να μπορέσει να ενισχύσει την επόμενη γενιά. γιατί δίνουμε μεγάλη έμφαση στο μέλλον. Όλα αυτά βεβαίως δεν μπορούν να γίνουν χωρίς ξεκάθαρες και ισχυρές εταιρικέ αξίες, όπως η αποδοχή της κοινωνικής ευθύνης. Και αυτό μας συνδέει άμεσα με τη νέα γενιά των παγκόσμιων μεταναστών, οι οποίοι προσελκύονται από την Deutsche Post, γιατί ακριβώς έχουν δυνατότητα να εισφέρουν στην ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον τελευταίο μιλητή και τους προηγούμενους βέβαια. Να πω δύο λόγια για να ξεκινήσει η συζήτηση. Να θίξω δύο σημεία που, δεν, που απήχαν από τη σημερινή συζήτηση όταν μιλάμε για τις αγορές εργασίας και την μετανάστευση. Ε, καταρχάς, ε, το πρώτο θέμα είναι η ποικιλομορφία αν κοιτάξετε ποια είναι η σημερινή αγορά εργασία, καταρχά τα ποσοστά ανεργία, α πούμε. Έχουμε μια τεράστια ποικιλία από το 14,4% στην ε, Ισπανία έως το 3% το Δεκέμβριο ε, του 2008 στην Ολλανδία. Και τα ποσοστά απασχόλησης των ε, γυναικών μέχρι το 2010 είναι 6% απασχολησιμότητα των γυναικών. Ίσως ε, θα είναι ο μόνος στόχος που θα υλοποιήσουμε αυτό το 2010. Από την άλλη έχουμε τη Σουηδία που έχουν φτάσει στο 73% της απασχολησιμότητας και άλλες χώρες που είναι χειρότερες βέβαια. Έχουμε τεράστιες διαφορές λοιπόν στην ε, σύνθεση και στην δομή των ε, αγορών εργασίας. Και αυτό έχει τεράστιες συνέπειες στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες και οι αγορές εργασίας αντιδρούν στις κρίσεις. Και επομένως τεράστιες συνέπειες στη σύνθεση και στη δομή του πληθυσμού των μεταναστών ε, μπορεί να το θεωρήσετε περίεργο, αλλά μόνο 4 στους 10 μετανάστες ε, έρχονται στην Ευρώπη για εργασία. Οι υπόλοιποι έρχονται για οικογενειακή επανένωση, για αναζήτηση ασύλου κτλ. αυτό το 4 στα 10% είναι παραπλανητικό. Γιατί στην Ισπανία, ας πούμε, στη χώρα μου, 9 στους 10 μετανάστες έρχονται για δουλειά. Ενώ στη Δανία, στη Γαλλία και στι σκανδιναβικέ χώρε σε γέννη, μόνο ένα στου δέκα έρχεται για δουλειά. Επομένω, το πώ θα διαχειριστούμε την μετανάστευση ε, τίθεται και με όρου κοινωνική ένταξη στι ε, ε σκανδιναβικέ χώρε. Ενώ σε εμά τίθεται με όρου αγορά εργασία. Και εμεί λοιπόν πρέπει να προσαρμόσουμε τι πολιτικέ μα σε αυτή την ε, ποικίλη πραγματικότητα. Ε, αυτό ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε. Πώς θα βρούμε δηλαδή μια κοινή πολιτική, μια κοινή στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη αυτή την ποικιλομορφία της κατάστασης. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να αναφέρω πολύ σύντομα είναι το θέμα της επίπτωσης της ε, σημερινής κρίσης στις μεταναστευτικές ροές. Δεν ξέρουμε την επίπτωση ακόμα, αλλά αυτό που ξέρουμε θα είναι σημαντικότατη η επίπτωση. Δεν θα υπάρχει καμία πτυχή της αγοράς εργασίας που δεν θα επηρεαστεί από την κρίση. Και σίγουρα και οι μετανάστες θα επηρεαστούν. Επομένως, με βάση την παρελθούσα εμπειρία και την κοινή λογική, τα πράγματα δεν φαίνονται και πολύ καλά για τους μετανάστες τρίτων χωρών. Γιατί αυτοί οι μετανάστες, μέσα στην ποικιλομορφία τους, ε, πλήττονται από ένα πρόβλημα έλλειψης ε, ειδικότητας και δεξιοτήτων. Και συχνά δεν ανήκουν ε, στους μηχανισμούς, θα συμμετέχουν στους μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας. Επομένως, θα έχουν ε, αβέβαιες θέσεις απασχόλησης, δεν θα προστατεύονται κοινωνικά και επομένως είναι οι πρώτοι που θα πληγούν από την οικονομική κρίση και την αυξανόμενη ενεργεία. Αυτή, αυτός ο προβληματισμός θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τη μετανάστευση. Και δύο-τρία τελευταία σχόλια. Για να συνοψίσουμε αυτά που ακούσαμε σήμερα, μου φέρνουν στο μυαλό το Max Fritz, έναν ελβετό συγγραφέα, Ελβετία που έχει τεράστια εμπειρία από τη μετανάστευση, ο οποίος τι είπε. Είπε ότι αυτό που θέλαμε ήταν όπλα, αλλά μας δόθηκαν άνθρωποι. Οι μετανάστες θεωρούνται, αντιμετωπίζονται ως εργατικό δυναμικό, ως ροές, αλλά είναι άνθρωποι. Περνάνε τα σύνορα και γίνονται πολίτες, γίνονται εργαζόμενοι. Η κυρία Κάν από την Νορβηγία πολύ σωστά είπε ότι αυτές οι χώρες που κατάφεραν να διαχειριστούν σωστά τη μετανάστευση είναι αυτοί που ένταξαν ε, τους μετανάστες, τους θεώρησαν τμήμα του εργατικού δυναμικού, τμήμα της κοινότητας που πρέπει να εντάξουν, όχι ως ε, τμήμα ε, της, ε, του εργατικού δυναμικού που θα πρέπει να το αναβοσβήνουν, να το προσαρμόσουν ας πούμε, ανάλογα με τι ανάγκε τη αγορά εργασία. Επομένω, θα πρέπει να διαχειριστούμε τη μετανάστευση με βιώσιμο τρόπο, με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, γιατί η μετανάστευση μα αρέσει ή δεν μα αρέσει, θα είναι μόνιμο στοιχείο τη κοινωνία μα για δημοκρατικού λόγου λόγω τη παγκοσμιοποίηση, γιατί ήδη είμαστε κοινωνίε ποικίλε και όχι μόνο σήμαντες. Θα πρέπει λοιπόν ε, με ευαισθησία, με ανθρωπιά ε, και με στρατηγικό όραμα να διαχειριστούμε τη μετανάστευση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα φύλλα, ε, το πρόβλημα της φυγής εγκεφάλων και το γεγονός ότι τελικά έχει σημασία το να έχει κανείς ειδίκευση και προσόντα. Τα προσόντα θα βοηθήσουν τους μετανάστες να ενταχθούν με υγιή τρόπο στην αγορά εργασίας. Διάφορες ερωτήσεις λοιπόν τέθηκαν και θα συμφωνήσετε όλοι ότι οι εμπειρογνώμονε του πάνελ έκαναν πολύ καλές παρουσιάσεις και τώρα έχετε εσεί το λόγο για να θέσετε τα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ πολύ τα μέλη του πάνελ το κύριο, και τον κύριο Πράτσιμον. Έχουμε αρκετό χρόνο για τη συζήτηση. Όσοι θέλουν να πάρουν το λόγο και δεν έχουν εγγραφεί μπορούν να σηκώσουν το χέρι. Θα τους δώσω το λόγο. Αλλά ο πρώτος ομιλητής είναι ένας Πολωνός γερουσιαστής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σε επιστήσω την προσοχή σε δύο προβλήματα. Τα οποία προέκυψαν από την παρέμβαση του Χαβιέρ Μονέ και των υπολείπων μελών του πάνελ. Το πρώτο θέμα είναι πόσο μακριά εμείς, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να πάμε σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση των πολιτικών μετανάστευσης. Εγώ είμαι νομικός, αυτό είναι το επάγγελμά μου, και μπορώ να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο νομικό επίπεδο έχει κάνει προσπάθειες για να εναρμονίσει τις νομικές της λύσεις, για να αντιμετωπίσει τους μετανάστες με εναρμονισμένο τρόπο, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους. Οι προηγούμενοι ομιλητές του πάνελ είπαν ότι το πρόβλημα της μετανάστευσης δεν έχουν να κάνουν με τις ανισότητες βορρά-νότου, αλλά και με τις ανισότητες ε, Ανατολής και Δύσης. Να μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύει τώρα πάνω σε δύο οδηγίες που θα εναρμονίσουν τις διαδικασίες χορήγησης ε, άδειας διαμονής και εργασίας για νόμιμους μετανάστες και νόμιμα διαμένονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η μία οδηγία. Η άλλη οδηγία, την οποία επεξεργαζόμαστε τώρα, είναι η οδηγία για τις προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μία γίνεται μια προσπάθεια εναρμόνισης και από την άλλη βέβαια πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο απέναντι σε αυτά τα θέματα. δεν προτιμάνε όλοι οι ξένοι μετανάστες το ίδιο όλες τις χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα, αν ένα Ευρωπαίο πολίτη θέλει μια δουλειά και ένα μετανάστη την ίδια δουλειά, θα πρέπει ο εργοδότη να δώσει προτεραιότητα στον ε, κοινοτικό πολίτη. Επίση, ένα άλλο θέμα είναι η αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών για να επιτρέψουν στου υπηκόου των χωρών να εισέλθουν στην αγορά εργασία. Επομένω, ποιο είναι το επίπεδο αυτονομία που έχει κάθε κράτος μέλος και σε, κάποιο, και σε ποιο βαθμό ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσπαθήσει να συντονίσει αυτές τις πολιτικές. Αυτές είναι πραγματικές προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κυρίε. Ε, υπάρχουν άλλα μέλη τα οποία θα ήθελα να παρέμβουν σε σχέση με κάποια από τα θέματα που αναπτύχθησαν εδώ. Κανείς δεν έχει κάποιο, κάποια ερώτηση, δεν θέλει να μας πει κάτι. Έχω μία ερώτηση για την κυρία Καν. Αν η Νορβηγία και οι σκανδιναβικές χώρες αλλάζουν τη μεταναστευτική τους πολιτική, από μια πολιτική που να μεταχειρίζεται τους εργαζόμενους σαν gastarbeiter, να τους αντιμετωπίζουν τώρα σαν μόνιμους πολίτες αυτής της χώρας. Ε, ποιο είναι το επίπεδο της συζήτησης στην Νορβηγία και στις άλλες σκανδιναβικές χώρες σε σχέση με τα ήθη της χώρας προορισμού ε, πώς γίνεται η ενσωμάτωση, πώς γίνεται η κατάρτιση της γλώσσας, Υπάρχει, υπάρχουν εξετάσεις στη γλώσσα ε, για να αποκτήσει κανείς την ηθαγένεια, πώς γίνεται κανείς ε, κανονικός πολίτης αυτής της χώρας αφορά τους παλαιούς μετανάστες, σε ποιους εφαρμόζονται, πώς εφαρμόζονται τα πρακτικά μέτρα αυτής της νέας πολιτικής. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντόντι. Κυρία, θέλατε να πάρετε το λόγο νομίζω. Ναι, ήθελα να πω κάποια πράγματα, γιατί εγώ ήδη είμαι μετανασ... μετανάστευσα στη Γαλλία και ήθελα να αναφερθώ στα όσα είπε η κυρία Καν για την Ορβηγία. Πιστεύω ότι εγώ ε, ε, στην περιοχή μας υπάρχει μια τοπική υπηρεσία στο Κροτέι, η οποία λειτουργούσε θαυμάσια και η οποία δεν είχε αρκετούς πόρους και την έκλεισαν. Λοιπόν, πάντοτε το πρόβλημα είναι το πώς θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά τα μέτρα. Ε, οι άνθρωποι γνωρίζουν πως πρέπει να επεξεργαστούν τα θέματα αυτά, όπως ο κύριος Γκαρσόν για παράδειγμα, ο οποίος είναι εξοικειωμένος με αυτά τα θέματα εδώ και πολλά χρόνια τα παιδιά των μεταναστών που είναι ε, ένα μελλοντικό δυναμικό. Δηλαδή, ε, εγώ έφτασα σε αυτή τη χώρα, αλλά δεν ισχύει για όλους αυτό. Ε, μπορεί κανείς να, να έχει μια υψηλή εξειδίκευση, να έχει υψηλά προσόντα. Υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι που έρχονται από τη Δυτική Αφρική ε, και που εκμεταλλεύονται ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες ε, χρηματοδοτούν σε αυτούς τους ανθρώπους. Εάν επενδύεται λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους και αν αυτή η επένδυση είναι εις των χωρών αυτών του Καναδά, λοιπόν, εδώ αναφύεται ένα πρόβλημα. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δίδεται μία εκπαίδευση στα στελέχη των υπηρεσιών αυτών όσον αφορά την ενίσχυση αυτών των ανθρώπων και την πρόθεση της σταδιοδρομίας τους. Γιατί ο μετανάστης με ποιον έρχεται σε επαφή, έρχεται πρώτα με, το, με τις τοπικές αρχές, με την κοινότητα. Θα πρέπει λοιπόν να ενεργοποιηθούν οι πόροι στο επίπεδο της κοινότητας, στο επίπεδο των δημοτικών αρχών γιατί εκεί φτάνουν τα προβλήματα. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής δεν ήταν έτσι διαμορφωμένη η πολιτική. Στο επίπεδο της Κομισιόν ισχύει το άρθρο 13 των συμφωνιών του Κοτονού. Είναι θέματα τα οποία έχουμε δουλέψει. Γιατί λοιπόν δεν εφαρμόζονται. Ε, θα πρέπει κάπως να προστεθούν οι διαδικασίες. Λέγονται πολλά λόγια, αλλά στο επίπεδο των ευρωπαϊκών διαδικασιών νομίζω εκεί υπάρχουν πολλά κενά ε, και θα πρέπει να γίνουν κάποιες προσπάθειες. Ο κύριος Λοζόν ζήτησε το λόγο και στη συνέχεια η κυρία Ζίλμπερτ Ρόμπερτς, ο κύριος Λοζόν. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι επικεφαλής της Λέσης για τις Σεϊχέλες ε, Δυτική Αφρική. Συνεργαζόμαστε με τον ΟΣΑ και δουλεύουμε συγγνώμη, με τη Σαχάρα. Ε, όταν μιλάμε για τη μετανάστευση πρέπει να λάβουμε υπόψη τα, τις δημογραφικές τάσεις και αυτό θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αν δούμε τις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε εμείς, ε, υπάρχει μια τεράστια αύξηση του πληθυσμού. Ε, η στρατηγική του 60 45 τώρα είναι 300 εκατομμύρια και το 2025 θα είναι 450 εκατομμύρια υπολογίστου. Δηλαδή δεν μιλάμε για ένα μικρό πληθυσμό. Δεύτερον, η δεύτερη πτυχή είναι ότι υπάρχουν 65% του πληθυσμού κάτω από, το 25, ε, κάτω από τα 25 όριο ηλικίας, ε, ηλικία. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τη Δυτική Αφρική, αλλά ισχύει και για το Μαγκρέπ και για τις υπόλοιπες αφρικανικές χώρες. Συνεπώς για μένα είναι δύο ερωτήματα σημαντικά όταν μιλούμε για τη μετανάστευση πού και πόσο θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι και ποιε είναι οι προοπτικές για την νεολαία. Όταν μιλάμε για την ανάπτυξη, πραγματικά θα πρέπει να ασχοληθούμε με το τι θα γίνει με την νεολαία. Γιατί οι νέοι αντιπροσωπεύει, όπω σα είπα, αντιπροσωπεύουν συγγνώμη, ένα τεράστιο τμήμα του πληθυσμού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λοζόν και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Τζίλμπετ Ρόμπερτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Διερωτώ μου τι μπορούμε να περιμένουμε όσον αφορά τη χρηματοοικονομική κρίση και τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. Την ποιότητα της αγοράς εργασίας. Ναι, συνήθως οι άνθρωποι μεταναστεύουν για μια καλύτερη ποιότητα ζωής κλπ. κλπ. Αλλά εν γέννη σε ένα πλαίσιο που πιστεύουν ότι είναι σε θέση να εισφέρουν και οι ίδιοι στην αγορά εργασίας, στη χώρα προορισμού. Θα μεταναστεύσουν ενδεχομένως περισσότεροι άνθρωποι ε, λόγω απελπισίας και δεν θα, φέρουν, θα έχουν συνεπώς αυτή την ποιότητα ε, στη νέα χώρα στην οποία έρχονται. Ίσως άνθρωποι με υψηλά προσόντα δεχομένω τώρα θα έχουν την αίσθηση ότι δεν θέλουν να διατρέξουν τον κίνδυνο, τους κινδύνους της μετανάστευσης. Ε, θέτω αυτό το ερώτημα, ίσως θα υπάρξει μια μετατόπιση που θα μας ε, υποχρεώσει να επανεξετάσουμε τους τρόπους διαχείρισης της αγοράς εργασίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κουνέλ, μέλος της Bundesrat από την Αυστρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω ορισμένες ερωτήσεις στο πλαίσιο αυτό. Πρώτον, οι χώρες που εκπροσωπούνται εδώ στο πάνελ έχουν αναπτύξει κάποιες ε, διαδικασίες ε, για να ε, διακρίνουν τους ετούντες άσυλο από τους οικονομικούς πρόσφυγες. Δεύτερον, έχετε προγράμματα εκπαίδευσης, γιατί ακούσαμε ότι σε ορισμένες ε, χώρες, ε, οι ενειδίκευτοι εργαζόμενοι δεν έχουν πολλά πράγματα να κάνουν. Αλλά υπάρχει μεγάλη ανάγκη ιδιαιτέρως ειδικευμένων εργαζόμενων. Και προσανατολίζεστε κυρίως σε αυτούς και όχι στους ανειδίκευτους. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν ξέχασα κανένα. Δεν θέλω κανένα να βγει από εδώ και να πει ότι ήθελε να μιλήσει και δεν τον είδα. Δεν θέλει κανένα να μιλήσει, βλέπω δεν σηκώνει κανένα το χέρι. Επομένω, τελειώσαμε τι ερωτήσει του κοινού. Ε, θα ήθελα ο κύριο Πράτ, ο συντονιστή, ο, ο κύριο Πράτ Μον, να οργανώσει την απάντηση. Θα δώσω το λόγο σε έναν έναν από τους εμπειρογνώμονες του πάνελ. Θα ξεκινήσω αντίστροφα από τον τρόπο με τον οποίο μίλησαν στην αρχή οι ομιλητές. Η κυρία Τζαμάικα πρώτη και καλύτερη. Ευχαριστώ. Από τα σχόλια που ακούστηκαν είναι προφανές ότι η μετανάστευση είναι μια δυναμική διαδικασία. Εξελίσσεται κάθε μέρα. Οι παγκόσμιες συνθήκες ούτως ή άλλως επηρεάζουν τα μοντέλα μετανάστευσης και τις φυγόκεντρες και κεντρομόλες τάσεις. Τι αναγκάζει κάποιον να φύγει και τι προσελκύει κάποιον ε, σε μια συγκεκριμένη χώρα. Ε, είναι πολύ επίκαιρη η συζήτηση βέβαια, δεδομένης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Επομένως, οι προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση είναι καταρχάς να προχωρήσουμε τη συζήτηση, να τη φτάσουμε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, εκεί όπου ε, προωθούνται οι πολιτικές και να βρούμε και κάποια κοινά θεμέλια πάνω στα οποία θα βασίσουμε τις ε, πολιτικές μας. Να υπάρξει μια συνοχή της μεταναστευτικής πολιτικής και να συνδεθεί με την ανάπτυξη. Εξελίσσεται λοιπόν αυτή η πολιτική, είναι, είναι μια δυναμική διαδικασία, επομένως δεν υπάρχει μία απάντηση που μπορούμε να δώσουμε τώρα. Πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τη διαδικασία και να δούμε αν υπάρχουν κάποιοι κοινοί παρανομαστές για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να εποφεληθούμε από τα πλεονεκτήματα και να μειώσουμε τα μειονεκτήματα. Να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων. Thank Um, Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση του κυρίου Ντάμπη. Βεβαίω πρέπει να κάνουμε ελκυστική στην Νορβηγία. Η Νορβηγία δεν είναι ελκυστική για όλους. Είναι πολύ ε, κρύα χώρα, έχει πολικές αρκούδες δίπλα στο Βόρειο Πόλο κτλ. Αλλά ο, ο, εκείνο που λέμε εμείς Εκείνο που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα για τους ξένους, για τους μετανάστες που έρχονται να δουλέψει είναι ε, το θέμα της ισότητας. Λέμε ότι πιστεύουμε στην ίση μεταχείριση, μιλάμε για την περίθαλψη, για την κοινωνική ασφάλιση, για την Ορβηγία από αυτή την άποψη πολύ πλούσια χώρα όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και προστασία. Όμως οι μετανάστες με τα πολλά προσόντα πάνε στον Καναδά και στις Ηνωμένε Πολιτείε οι άντε να πάνε και στη Μεγάλη Βρετανία δεν έχουμε ε, δεν έρχονται στην Νορβηγία Οπότε αναρωτιέται κανείς έστω ότι έρθουν ας πούμε γιατί σε εμάς έρχονται από την Ασία, από την Ινδία και τα λοιπά ε, όπως είπαμε ε, το ερώτημα είναι μήπως εμείς δημιουργούμε ουσιαστικά τη διαρροή εγκεφάλων από τις χώρες της Ασίας μπαίνει ένα ισκό πρόβλημα πλέον εκεί τώρα τι ε, καταλαβαίνουμε από τους δικούς μας τους κανόνες και από δική μας την κοινωνία η μετανάστες. Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσουμε το ερώτημα. η μετανάστες πολύ διαφορετική εμείς όταν συζητάμε την μετανάστευση και τους ε, ετούντες άσυλο και θέματα επανένωσης οικογενειών κτλ. Μιλάμε γενικώ για μετανάστες σαν όλοι οι μετανάστες να είναι ίδιοι. Ε, αυτό είναι λάθος και είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που, που κάνουμε αυτό διότι εδώ μιλάμε για μετανάστες από τη μια πρόσφυγες από την άλλη λαθρομετανάστες μουσουλμάνους ε, ε Εβραίους, Καθολικούς, Άθεους. Τι να σας πω, υπάρχουν πάρα, πάρα πολλές κατηγορίες ε, μεταναστών ε, ε, και οι διαφορές μεταξύ των κατηγοριών αυτών είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι μεταξύ των του Αμερικανού από το Κολοράντο και του από την Καλιφόρνια και από τη Νέα Υόρκη ας πούμε τέλος πάντων είναι πολύ πολύ δύσκολο να ε, δούμε και από κοινού όλους τους μετανάστες η γυναίκα από τη Σομαλία που είναι αναλφάβητη δεν έρχεται δεν ήθελε να έρθει στην Νορβηγία αλλά δεν είχε καμιά άλλη επιλογή έπρεπε να ακολουθήσει τον άντρα της ο οποίος άντρας επίσης δεν ήθελε να έρθει στην Νορβηγία αλλά δεν έχει δουλειά ή δεν μπορεί να επιβιώσει την κοινωνία από την οποία έρχεται ε, Θα είμαι πολύ σύντομος στην, ε, στις καλύτερες, ε, στην καλύτερη περίπτωση που θα υπάρχει αναδιονομή του πλούτου στον κόσμο θα αριθμιστούν οι μεταναστευτικές ε, ροές. Παρόλα αυτά θα συνεχίσουν, ακόμα και αν υπάρχει αναδιανομή του πλούτου. Συνεπώς, αυτό το οποίο είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα προϋποθέτει μια παγκόσμια λύση, παγκόσμιους κανόνες και παγκόσμιους θεσμούς που να τη ρυθμίζουν. Όσον αφορά την ερώτηση για το βαθμό εναρμόνισης που πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στη μετανάστευση, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είμαι ειδικό για να απαντήσω αυτή την ερώτηση, γιατί έχω μόνο δέκα μήνες σε αυτό το κοινοβούλιο και αυτούς τους δέκα μήνες ακόμα ε, δεν είχα το χρόνο να ε, μελετήσω διαφορετικά συστήματα που ισχύουν στην Ευρώπη. Σε συνάρτηση με το όραμα της Ευρώπης που θέλουμε να έχουμε θα πρέπει να γίνει και η εναρμόνιση της μεταναστευτικής πολιτικής. Ε, μιλάμε για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν έχει ακόμα επιτευχθεί εναρμόνιση. Συνεπώς, ε, η επίλυση που ζητάμε όσον αφορά την εναρμόνιση της μετανάστευσης είναι κάτι το οποίο, για το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε πολύ. Βεβαίως ε, έχει δοθεί μία όθηση στην κατεύθυνση αυτή και μπορούμε στο μέλλον να εμβαθύνουμε πολύ περισσότερο. Παρακαλώ να χρησιμοποιήσουμε τα υπόλοιπα λεπτά για να εμβαθύνουμε στα ερωτήματα. Υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης εναρμόνισης. Ναι. Ε, Κοιτάξτε, εκείνο που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να δούμε όλες τις εθνικές νομοθεσίες για να δούμε τι είναι ε, εφικτό και τι δεν είναι. Ε, αν τελικά δούμε ότι το άλλο ερώτημα τώρα είναι αν πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε η positive discrimination ε, είναι η θετική διάκριση για να προωθηθούν κάποιες κατηγορίες οι οποίες μέχρι τώρα έχουν αδικηθεί δεν ξέρω ε, Τώρα για τους μετανάστες περιμένουμε να υπάρξει κάποιο κέρδος από αυτούς ή να αποδώσει η επένδυσή μας αν θέλετε στο μετανάστη. Ναι, όντως ε, μπορούμε να φανταστούμε ότι θα υπάρξει κάποια, κάποιο κέρδος από την επένδυση αυτή αλλά σε πολύ γενικούς όρους ίσως όχι ποσοτικά εκφραζόμενους ε, από εκεί και πέρα ε, για την ε, κοινωνική ασφάλεια και προστασία ε, τι να σας πω, δεν ξέρω, κάποιες κυβερνήσεις ανέλαβαν ε, κάποιες πρωτοβουλίες ή είπαν ότι παίρνουν κάποια μέτρα. Ε, εμείς σαν εταιρεία δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Αλλά το επόμενο ερώτημα που έχω σημειώσει εδώ, αν επηρεάζεται η αγορά εργασίας από την ε, μετανάστευση, μα βεβαίως δεν υπάρχει, συμβαίνουν πάρα πολλά παράξενα πράγματα στην αγορά εργασίας παντού ε, αυτή τη στιγμή ε, και η σχέση με τη μαφία είναι κάτι που δεν το βλέπει κανείς μόνο στις κινηματογραφικές ταινίες. ίσως είναι και πραγματικότητα οι μαφίες εντός εισαγωγικών η... είναι σημαντικό να καθίσουμε να σκεφτούμε ότι η λαθρομετανάστευση όπως και να την ονομάσουμε τώρα μπορεί να μοιάζει και μοιάζει σε πολλές περιπτώσεις με το παλιό σκλαβεμπόριο τώρα Israel and the animation. Ε, αν δει κανείς ε, αν ε, δει κανεί ε, τώρα πώ μπορεί εν πάση περιπτώσει να κερδίσει και χώρα προέλευση από κάποια πράγματα ε, κοιτάξτε διαφημίσει, παραδείγματο χάρη όπου το, το, το γύρισμα γίνεται στην Ταϊλάνδη το, το, μοντάζ σε μια άλλη ασιατική χώρα κτλ. κτλ. Αυτός είναι ένας τρόπο να επανέλθουν τα κέρδη στη χώρα προέλευση, αν θέλετε. Και τώρα Ο λόγος στον κύριο Ζακ Μπαγό, επίτροπο υπεύθυνο για θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, ε, υπεύθυνος για θέματα ασύλου και μετανάστευση είναι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τη στιγμή που ανέλαβε αυτά καθήκοντα ε, στα μέσα του 2008 ε, ασχολήθηκε πραγματικά με ζήλο και έδωσε μια νέα διάσταση σε αυτές τις πολιτικές. Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Ντεπρέ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους όσους μίλησαν σε αυτή την κοινοβουλευτική διάσκεψη για την συνέπεια και συνοχή των πολιτικών ανάπτυξης και της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Δουλέψατε πολύ καλά. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα αποτέλεσμα από αυτή την προσπάθεια που κάνατε, από τις συνεισφορές σας, από τις παρεμβάσεις σας. Ε, μια πολύ σημαντική στιγμή για μας, γιατί θα πρέπει λίγο-λίγο να εφαρμόσω αυτή την πολιτική, η οποία αποτελεί αντικείμενο συνένεσης γύρω από το σύμφωνο ε, μετανάστευσης και ασύλου που υιοθετήθηκε επί Γαλλικής Προεδρίας. Τώρα, το 2009 θα προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε την πολιτική ασύλου και εν συνεχεία βεβαίως θα πρέπει να αναπτύξουμε την, ε, μια πολιτική σφαιρική για να συνδέσουμε τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών με την ανάπτυξη. Θα σας μιλήσω για αυτό σε λίγο. Φυσικά είμαστε βυθισμένοι σε μια οικονομική κρίση που πλήττει κατά μέτωπο τις οικονομίες μας ε, και των, ε, τις δικές μας και των εταίρων μας και θα είναι πολύ πιο δύσκολο κατά τη διάρκεια της κρίσης να διαχειριστούμε τις μεταναστευτικές ροές. αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες μας. Θα πρέπει να δούμε οι αποφάσεις μας, ε, τι επιπτώσεις θα έχουν στην ισορροπία των κοινωνιών μας, των κοινωνιών των εταίρων μας και η ανάπτυξη επίσης των εταίρων μας. Γιατί μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη αυτών που μας στέλνουν μετανάστες. Μια και δεν υπάρχει ανάπτυξη στις χώρες τους, είναι αναγκασμένοι λοιπόν να φύγουν από εκεί και να μεταναστεύσουν. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για αυτή την σφαιρική προσέγγιση. Οι δεξιότητες και τα προσόντα που έχουν συλλέξει οι μετανάστες στην εμπειρία τους στο εξωτερικό μπορούν να γίνουν μοχλή σημαντική για την ανάπτυξη. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να έχουν αυτή την ευκαιρία η σχέση μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης αποτέλεσε αντικείμενο πολλών παρεμβάσεων και προβληματισμών και συζητήσεων φυσικά ε, σε ό,τι αφορά τη συνεισφορά της διασποράς στην ανάπτυξη της χώρας προέλευσης και σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των κονδυλίων και σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της διαρροής των εγκεφάλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να εντάξει καλύτερα αυτή τη διάσταση των μεταναστευτικών ροών στην πολιτική της εξωτερικών σχέσεων, απασχόλησης, τις οικονομικές πολιτικές, πολιτικές υγείας και κοινωνικών υποθέσεων. Το 2008, υπενθυμίζω, ήταν μια ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Αυτό το σύμφωνο ε, έχει τις βασικές αρχές της κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο. Η σφαιρική προσέγγιση της μετανάστευσης βασίζεται σε μια ισορροπημένη μεταχείριση των διαφόρων πτυχών της μετανάστευσης. Θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι τώρα σε αυτό το σημείο. Αυτή, αυτό το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο δεν διέπεται από μια λογική που έχει να κάνει μόνο με την ασφάλεια. Φυσικά θα πρέπει να προλάβουμε και να μειώσουμε τη λαθρομετανάστευση. Γιατί η λαθρομετανάστευση οργανώνεται κυρίως από ενδιάμεσους οι οποίοι συνδέονται με κάποιο τρόπο με το οργανωμένο έγκλημα. Ε, έχουμε λοιπόν καθήκον να καταπολεμήσουμε την λαθρομετανάστευση. Αλλά δεν τελειώνει εδώ η σφαιρική προσέγγιση. Παράλληλα, θα πρέπει να οργανώσουμε και να διαχειριστούμε την νόμιμη μετανάστευση. Θα πρέπει να προστατεύσουμε του μετανάστε που είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνου εμπορία, εκμετάλλευση και ρατσισμού. Θα πρέπει να προωθήσουμε τα δικαιώματα των προσφύγων και όσων χρήζουν προστασίας. Η σφαιρική προσέγγιση σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενσωματώσει την ε, μεταναστευτική πολιτική στις αναπτυξιακές πολιτικές για να δούμε πώς ε, οι πολιτικές αυτές μπορούν να βοηθήσουν τις χώρες προέλευσης. Με αυτή την ε, σφαιρική προσέγγιση θέλουμε να δημιουργήσουμε πολιτικούς και θεσμικούς μηχανισμούς που θα μας επιτρέψουν να διαχειριστούμε με συνεπή τρόπο και ισορροπημένο τρόπο την μετανάστευση μαζί με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες με σεβασμό της δικής τους ανάπτυξης. Ακριβώς γι' αυτό εγώ προσωπικά τόνισα ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον εξή όρο. Μια συντονισμένη διαχείριση της μετανάστευσης και των μεταναστευτικών ροών. Συντονισμός. Δεν μπορεί να διαχειριστούμε μακροπρόθεσμα τη μετανάστευση χωρίς να έχουμε διάλογο και μάλιστα συνεχή διάλογο με τις χώρες προέλευσης. Να πώς θα τα καταφέρουμε να ενσωματώσουμε την αναπτυξιακή πολιτική και τη μεταναστευτική πολιτική. Θα μιλήσω τώρα για συγκεκριμένα πράγματα όπου προσπαθούμε πραγματικά να υλοποιήσουμε αυτή τη σφαιρική προσέγγιση. Τα πέντε τελευταία χρόνια η κοινότητα ε, χρηματοδότησε πάνω από 150 προγράμματα συνεργασίας με τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης. Ε, πρόσφατα δρομολόγησα συνεργασία μαζί με το πρόγραμμα του ΟΗΕ για την ανάπτυξη, μια πρωτοβουλία με 15 εκατομμύρια ευρώ με στόχο να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο για τις τοπικές αρχές και τις οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών, των κρατών μελών και 15 τρίτων χωρών, ούτως ώστε να προωθήσουμε την τοπική ανάπτυξη μέσω της κινητοποίησης των κοινοτήτων των μεταναστών. Στην Κάναγα, στο Σαλβαντόρ, στις Φιλιππίνες, στο Μαρόκο, η Κομισιόν, σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προσπαθεί να διευκολύνει την μεταφορά των κονδυλίων των μεταναστών να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια για χρήσιμε χρήσιμες πρωτοβουλίες στις χώρες προέλευσης. Τρίτο παράδειγμα, δημιουργήσαμε την εταιρική σχέση για την κινητικότητα με τη Μολδαβία και το Πράσινο Κροτήρι. Σε αυτά τα προγράμματα εταιρική σχέσης προσπαθούμε να εντάξουμε επαγγελματικά και κοινωνικά τα άτομα που επιστρέφουν. Σε αυτές τις συμφωνίες εταιρική σχέση υπάρχουν και συμφωνίες επανεισδοχής που φυσικά επιτρέπουν να στείλουμε πίσω τους λαθρομετανάστες αλλά να τους εξασφαλίσουμε παράλληλα κατά την επιστροφή τους έτσι, μια πλαισίωση Παράλληλα, αυτές οι συμφωνίες, οι οποίες είναι παραδειγματικές, επιτρέπουν να συμμετάσχουμε εμείς σε αναπτυξιακές ε, δράσεις. Τέταρτον, έχουμε πιλωτικές πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά την κυκλική μετανάστευση. Η κυκλική μετανάστευση σημαίνει ότι είναι προσωρινή μετανάθεση προς την Ένωση ή προσωρινή επιστροφή των ειδικευμένων με σκοπό να μεταφέρουν τις γνώσεις τους ή να δουλέψουν για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της χώρας τους. Όταν, και εδώ ευχαριστώ τον πρόεδρο Ντεπρέ, ο οποίος μας βοήθησε να υλοποιήσουμε το πρώτο βήμα της Μπλε Χάρτα χάρτας που επιτρέπουν στους ειδικευμένους εργαζόμενους να έρθουν να δουλέψουν στην Ευρώπη μέσα σε πιο ελκυστικές συνθήκες και σε λίγες εβδομάδες θα παρουσιάσω ένα κείμενο για τους εποχιακούς εργαζόμενους, για τους μαθητευόμενους που πληρώνονται. Μέσα από αυτά τα κείμενα προσπαθούμε να υλοποιήσουμε την κυκλική μετανάστευση. Θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι που έρχονται στην Ευρώπη να μπορούν εν συνεχεία να επιστρέψουν στη χώρα πρόληψής τους και να εποφεληθούν οι συμπατριώτες τους από την εμπειρία τους στο εξωτερικό. Επίσης, συνεισφέραμε τα τελευταία χρόνια για την εφαρμογή κέντρων για την κατάρτιση και τη διαχείριση της μετανάστευσης. Τα κέντρα αυτά συμβουλεύουν τους ενδεχόμενους υποψήφιους για τη μετανάστευση, αλλά και καταρτίζουν ή προσανατολίζουν τους μετανάστες προς συγκεκριμένους προορισμούς. Έχουμε πράγματος χάρη στο Μαρόκο, ε, την ΑΠΕΚ, το ΣΥΖΕΜ που μόλις ξεκίνησε στο Μαλί και επίσης θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε ε, και να προωθήσουμε αυτή την ενημέρωση των υποψηφίων για τη μετανάστευση στις χώρες προέλευσης. Αυτά είναι απλώς κάποια παραδείγματα. Θέλω να σας πω, δεν υπάρχει διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αν υπάρχει στενή συνεργασία με τις χώρες προέλευσης. Αυτό είναι προϋπόθεση. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και υπομονή. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μία διαπραγμάτευση με την Σενεγάλη, μία άλλη με το Μαρόκο, Δεν είναι εύκολες αυτές οι διαπραγματεύσει, γιατί φυσικά θέλουμε να υπάρξουν και συμφωνίε επανεισδοχή για τους λάθρομετανάστες. Αλλά βεβαίω θέλουμε σαν αντιστάθμισμα να δώσουμε και κάποια βοήθεια. Φυσικά, αυτές οι χώρες μας λένε πολύ ωραία να υπογράψουμε συμφωνίες επανεισδοχής για τους δικούς μας υπηκόους, αλλά επειδή είμαστε και χώρες διαμετακόμισης είναι δύσκολο. Τι θέλω να σας πω, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ας με διορθώσει αν κάνω λάθος ο πρόεδρος της ε, πιο αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, ο κ. Ντεπρέ, πιστεύω λοιπόν ότι θα ήταν λάθος για τη μεταναστευτική μας πολιτική να την αντιμετωπίσουμε από την σκοπιά της ε, ασφάλειας, ε, να προστατεύσουμε τις αγορές εργασίας να επιλέξουμε τους μετανάστες ανάλογα με τις ανάγκες μας χωρίς να δίνουμε καμία σημασία στις ανάγκες των χωρών προέλευσης. Χρειάστηκε μετά από την οδηγία για τις επαναπροωθήσεις να εξηγήσω ειδικά στη Λατινική Αμερική ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η οδηγία για τις ε, επιστροφές δεν είναι τέλεια, είναι ένα πρώτο βήμα. Μας επιτρέπει να έχουμε ένα νομικό πλαίσιο για να οργανώσουμε κάπως καλύτερα τις επιστροφές της, τον επαναπατρισμό των ανθρώπων αυτών. Ε, παράλληλα, ε, έχουμε και κείμενα για την ε, νόμιμη μετανάστευση και με αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε ένα σημείο ισορροπίας. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ευχαριστώ τον ΩΣΑ. Νομίζω ότι πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι οι φορείς, θα πρέπει να είμαστε συντονισμένοι σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές πολιτικές. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, διακυβεύονται πολλά. Θα πρέπει να μεταφέρουμε ε, τα κονδύλια, τα, τα, τα, τα κεφάλαια των μεταναστών προς τις χώρες προέλευσης με σκοπό την ανάπτυξη. Γιατί οι κοινότητες προέλευσης που παίρνουν αυτά τα κονδύλια θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικές τραπεζικές υπηρεσίες. Αυτό τι σημαίνει σε χώρες θα πρέπει να αναθεωρηθεί το τραπεζικό σύστημα. Παράλληλα είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ούτω ώστε μια μαζική μετανάστευση ε, επαγγελματιών της υγείας, ας πούμε, οδηγήσει στο να μην υπάρχουν γιατροί και νοσοκόμες στις ε, χώρες πρόεδρες. Θα πρέπει λοιπόν οι προσλήψεις εδώ να γίνονται με διοντολογικό τρόπο. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε τις τρίτες χώρες να μεταρρυθμίσουν τον τομέα της υγείας, ούτως ώστε αυτοί οι επαγγελματίες της υγείας να παραμένουν στις χώρες αυτές, γιατί έχουν ρόλο εκεί να παίξουν. Κάναμε πολύ πρόοδο για να έχουμε ένα συνεπές πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής με σκοπό την ανάπτυξη. Αλλά τα πιο δύσκολα δεν έχουν γίνει. Θα πρέπει να κινητοποιηθούμε εμείς, να κινητοποιήσουμε τους πόρους μας και θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε μια νέα κουλτούρα στην Ευρώπη, μια νέα αντίληψη για τη μεταναστευτική πολιτική. Μια κουλτούρα πολύ πιο ανοιχτή, παράλληλα όμως θα πρέπει να γίνει αυτό με κανόνες, κοινούς κανόνες, συντονισμένους κανόνες. Και επιμένως θα πρέπει να υπάρξει κέρδος και για μας και για τις χώρες προέλευσης. Θα πρέπει και εμείς και οι χώρες αυτές να επωφεληθούμε από αυτή τη διαχείριση της μετανάστευσης. Τους επόμενους μήνες θα γίνουμε μάρτυρες σε μεταναστευτικά φαινόμενα πολύ πιο έντονα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μετασχηματίσουμε αυτές, αυτά τα κύματα μετανάστευσης σε μετανάστευση έτσι επιλεγμένη, συντονισμένη. Εμείς δηλαδή, η Ευρώπη μαζί με τις ίδιες χώρες. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουμε ένα μοντέλο στην Ευρώπη, θα αποτελέσουμε στην Ευρώπη ένα μοντέλο διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής για αυτά τα αποτελέσματα που χαρακτηρίζονται από μέτρο, γιατί μιλάμε για ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο θέμα, που χαρακτηρίζονται από μια διάβια σε σχέση με το τι μας αναμένει στο μέλλον και από κουράγιο για όσον αφορά ε, την παρουσίαση των απόψεώς μας σε μια κοινή γνώμη η οποία δεν έχει πάντοτε επίγνωση του μεγέθους των προβλήματων και των προκλήσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές αυτής της διάσκεψης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον ΩΣΑ και την Επιτροπή. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια πρώτη συνδιάσκεψη αυτής της μορφής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς. Να ευχαριστήσω το σύνολο των συμμετεχόντων, του πάνελ και εσάς. Και εάν θέλετε να μας ξαναδείτε, να πάτε στο site του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και στην ιστοσελίδα web του ΟΟΣΑ. Ευχαριστώ πολύ.